Mes chers collègues, nous allons pouvoir commencer notre euh, séance, s'il vous plaît. Le projet d'ordre du jour, M. Marinescu et M. Kramer. Ας ξεκινήσουμε. Παρακαλώ πολύ πάρτε τις θέσεις σας. Το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης μπορεί να υιοθετηθεί αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Ε, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 10ης και 29ης Ιανουαρίου είναι διαθέσιμα. Μπορούμε να τα εγκρίνουμε αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Δεν έχω καμία ανακοίνωση. Τυχεράκιδες. Και έχω την τιμή να καλωσορίσω τον Ρουμάνο Υπουργό Τουρισμού Κύριε Υπουργέ, καλώ ήρθατε. Από την 1η Ιανουαρίου η Ρουμανία έχει αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου με πολλά φιλόδοξα σχέδια για το μέλλον της, Ευρω... της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον τομέα του τουρισμού. Όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα της Προεδρίας, ο τουρισμός αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και θα πρέπει να είναι πολύ πιο ορατός στην στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να, να δώσουμε μια ιδιαίτερη προσοχή στην, ε, στα μέτρα που έχουν ως στόχο ο τομέας αυτός να ενταχθεί περισσότερο στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος είναι ο τουρισμός να είναι βιώσιμος, υπεύθυνο, να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, κάτι που θα δώσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις μας, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπω επίση και στους Ευρωπαίους καταναλωτές στο σύνολό τους. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω κύριε Υπουργέ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι πάντα στην πρωτοπορία της ευρωπαϊκής πολιτικής τουρισμού. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την απόδοση ενός προπολογισμού όλο και πιο σημαντικού στο πλαίσιο του βιώσιμου τουρισμού στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2001-2027 δεδομένου ότι ο τουρισμός αποτελεί ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας στο σύνολό της. Έχουμε πολλά κοινά ενδιαφέροντα και πολλούς κοινού στόχους. Οπότε μπορείτε να βασιστείτε στην συνεργασία μας κύριε Υπουργέ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στην Προεδρία σας. Θα σας δώσω το λόγο για 10 περίπου λεπτά και μετά θα προχωρήσουμε σε μια ανταλλαγή απόψεων με τους ευρωβουλευτές. Καλώς ήρθατε. Stimată doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European,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 Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν λοιπόν ξεκινήσω θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι σας υποστηρίζω ανεπιφύλακτα γιατί έχουμε ένα κοινό στόχο συγκεκριμένα να προάγουμε τον τουρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πρώτος ε, στόχος των τουριστών και γι' αυτό πρέπει να συνεργαστούμε. Το 2018 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τον τουρισμό ο οποίος διευρύνθηκε στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στατιστικά δεδομένα που έχουμε καταδεικνύουν τις δυνατότητες που έχει ο τουρισμός ε, να ε, αναζωογονήσει την οικονομία, αλλά χρειαζόμαστε μια στρατηγική η οποία θα βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα. Για να γίνει όμως αυτό, χρειαζόμαστε γνώσεις ε, για τις προεκτάσεις του τουρισμού, ο οποίος είναι ένας δυναμικός τομέας, ο οποίος βέβαια υφίσταται συνεχείς αλλαγές. Παράλληλα, ο τουρισμό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη τη οικονομία με τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Αυτό λοιπόν είναι ένα επιπρόσθετο λόγο γιατί η πολιτική τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στεφτεί από επιτυχία. Τη χρειαζόμαστε αυτή την πολιτική έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί ένα ποιοτικό ε, στόχο και βιώσιμο στόχο των τουριστών. Και για να επιτευχθεί αυτό χρειαζόμαστε έναν πολιτικά φιλόδοξο στόχο. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη οφείλουν από κοινού να λάβουν και να εφαρμόσουν εφαρμόσουν μέτρα έτσι ώστε να διαφυλαχθεί η πολιτιστική κληρονομιά. Στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο προβλέπονται συγκεκριμένα προγράμματα και για στην κοινή αγορά προβλέπονται προγράμματα. Υπάρχει κατρεχόν καταρχά η πρόταση για τον κανονισμό σχετικά με τον τουρισμό όπου θα ρυθμιστούν η ανταγωνιστικότητα και η σταθεροποίηση των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Το ίδιο ισχύει και για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. <coughs> Όμως, για να ευθυγραμμιστεί η νομοθεσία, αυτές όλες οι ε, διατάξεις και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες πρέπει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Και για το λόγο αυτό χρειαζόμαστε επιπρόσθετες προσπάθειες. Γιατί μόνο έτσι έτσι μπορεί ο τουρισμός ε, να βρίσκεται στην αιχμή του δώρατος της, ε, του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου και να επιφέρει ανάπτυξη και απασχόληση. <clears throat> Ανάπτυξη λοιπόν ή μάλλον απασχόληση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο όπου ο κλάδος ε, διαμαρτύρεται ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Ο τουρισμός βέβαια υφίσταται τις εποχικές ε, μεταβολές και γι' αυτό τα πράγματα δυσχεραίνουν. Το φαινόμενο αυτό διαπιστώνεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα λοιπόν με τα μέτρα εκπαίδευσης που θα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε εκείνες τις πρωτοβουλίες ε, που οδηγούν στο να αυξηθεί η ε, δραστηριοποίηση στον τουρισμό. Το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε και μακροπρόθεσμα. Όπως σας είπα ήδη, Υπάρχει λοιπόν η βιωσιμότητα στον τουρισμό, η οποία είναι σε άμεση συνάρτηση των ε, εποχικών μεταβολών. Η Ρουμανία έχει θέσει ως στόχο να συνεχίσει την πορεία της Έχουμε λοιπόν ε, στο Συμβούλιο καταθέσει συγκεκριμένε προτάσει. Ε, θέλουμε να απευθυνθούμε σε συγκεκριμένα θέματα, ψηφιοποίηση, βιωσιμότητα, ε, συνεργασίες, εποχικότητα, κλιματική αλλαγή, υπερπληθώρα τουριστών σε κάποιους ε, αγαπημένους τουριστικούς ε, προορισμούς. Όπως σας είπα, τα κράτη-μέλη πρέπει να στηρίξουν την νοσιακή στρατηγική. Από κοινού λοιπόν με τα κράτη-μέλη οφείλουμε <clears throat> να αναζητήσουμε ένα στρατηγικό έγγραφο το οποίο θα περιλαμβάνει την ανακοίνωση της, ε, θα αντικαταστήσει μάλλον την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2010 και θα δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο για την ευρωπαϊκή πολιτική τουρισμού. Όλα αυτά θα πρέπει να προσαρμοστούν στην ψηφιοποίηση και στην κοινή αγορά και αυτά επιθυμούμε να τα συζητήσουμε ε, τέλος του έτους ε, στο Συμβούλιο που θα ασχοληθεί με θέματα ανταγωνισμού. Τουρισμός χωρίς νέες τεχνολογίες δεν μπορεί να υπάρχει. Τούτο λοιπόν απαιτεί να προσαρμοστούμε στη νέα ψηφιακή οικονομία. Και αυτό ισχύει προφανώς για όλους τους ε, τουριστικούς ε, προορισμούς. Για να μπορέσουμε να απολαύσουμε τα πλεονεκτήματα που μας προσφέρει η τεχνολογία, χρειαζόμαστε συγκεκριμένη πολιτική προσέγγιση, χρειαζόμαστε προγράμματα και χρειαζόμαστε και ένα θετικό επενδυτικό κλίμα για τις ε, επιχειρήσεις. Εδώ παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο οι νεόφυτες επιχειρήσεις, η εκβιομηχάνηση έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και γι' αυτό πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες τεχνολογίες. Και προς αυτή την κατεύθυνση χρειαζόμαστε την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι ε, νεόφυτες επιχειρήσεις βρίσκονται στο πυρήνα των προσπαθειών μας. Ε, Βεβαίως ε, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να εντοπιστούν οι ανάγκες ε, των νεόφυτων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην αρχή όλες οι επιχειρήσεις χρειάζονται βοήθεια, αλλά η βοήθεια αυτή δεν είναι παντού ίδια, ποικίλει. Ε, Γι' αυτό χρειαζόμαστε και μία προσαρμοσμένη πολιτική, προσφέρουμε, να προσφέρουμε τη δυνατότητα να αναπτυχθούν επιχειρήσεις. Υπάρχουν και συγκεκριμένα επιχειρηματικά μοντέλα. Παραδείγματος χάρη online πλατφόρμες, μέσω των οποίων μπορεί κανείς να υπενικιάσει ένα δωμάτιο στο ίδιο του το σπίτι. Αυτό βεβαίως και έχει επιπτώσει στον κλάδο και αυτή η διάσταση του προβλήματος δεν πρέπει να παραμελείται. Είναι σημαντική για τους ε, εμπειρογνώμενες του τόμου ε, του, του χώρου των ακινήτων. Ε, πρέπει να αποφύγουμε επίση ή δυνατόν ορισμένοι προορισμοί ε, να είναι υπερκαλυμμένοι. Βεβαίω χρειαζόμαστε υψηλέ προδιαγραφέ ποιότητα, αλλά χρειαζόμαστε και την προστασία των γηγενών. Υπάρχουν παρεμφερείς κλάδοι, ο πολιτιστικός κλάδος, ο δημιουργικό κλάδος. Πρέπει να υπάρχουν συνεργασίε ανάμεσα σε ΜΚΟ, ε, και ε, ιδιώτες επενδυτές. Και αυτό το μοντέλο μπορεί να επεκταθεί μόνο αν αποδώσουμε σημασία στην ποιότητα, έτσι ώστε οι τουριστικοί προορισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βρίσκονται στην ε, πρώτη βαθμίδα. Χρειαζόμαστε και καλύτερη ενσωμάτωση του τουρισμού στις πολιτικές προσπάθειες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βιωσιμότητα, υψηλή ποιότητα, αυτές είναι οι λέξεις κλειδί. Και Αργότερα αυτά αποδεικνύονται ως πλεονεκτήματα στην ανταγωνιστικότητα, τόσο για τις μικρομέσες επιχειρήσεις όσο και για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Όλα αυτά μπορούν να σημαίνουν πλεονεκτήματα. Χρειαζόμαστε ε, βιώσιμο τουρισμό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε ένα ευφυές πλαίσιο. Η βιωσιμότητα μακροπρόθεσμα χρειάζεται τη συνεργασία με τον τομέα του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και άλλους συναφείς τομείς. Παράλληλα υπάρχει και μια ηθική διάσταση του θέματος. Δηλαδή εμείς δεν επιθυμούμε ε, να υπάρξει, όπως σας είπα, υπερπληθώρα τουριστών σε κάποιους ε, τουριστικούς ε, προορισμούς. Θέλουμε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Αυτό λοιπόν σημαίνει κινητικότητα, διασύνδεση ανάμεσα στους προορισμούς και επίσης κάλυψη των αναγκών των ντόπιων πολιτών. Πράγματι, πρέπει να τηρήσω το χρόνο που μου έχετε διαθέσει και γι' αυτό και μίλησα πάρα πολύ γρήγορα. Η ε, ενότητα του τουρισμού πρέπει για όλους μας να είναι στόχος. Ως εκ τούτου ε, θα πρέπει να λάβουμε μέτρα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε ε, το πρόβλημα της ε, υπερπληθώρας τουριστών όπως σας ανέφερα. Γιατί αυτοί οι τουριστικοί προορισμοί εξακολουθούν να είναι χώρες, πόλεις όπου οι άνθρωποι εξακολουθούν να εργάζονται και θέλουν και αυτοί να διασκεδάζουν. Ο βιώσιμος τουρισμός είναι όπως σας είπα λέξη κλειδί. Παράλληλα ε, μπορούν να αναπτυχθούν και άλλες περιοχές μιας χώρας. Για να το πετύχουμε όμως αυτό, χρειαζόμαστε μια κοινή βάση δεδομένων. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να προάγουμε μόνο τους γνωστούς ε, τουριστικούς προορισμούς μέσω της διαφήμισης. Ε, πρέπει να επεκταθούμε και σε άλλες περιοχές. Υπάρχουν πολύ όμορφες περιοχές οι οποίες δεν είναι ακόμα τόσο γνωστές. Η υπερκάλυψη μπορεί να εκλειφθεί ως ένα κριτήριο. Ε, το κριτήριο αυτό θα πρέπει να είναι μεγάλη σημασία, να εξεταστεί για όλους αυτούς τους λόγους χρειαζόμαστε συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης, το οποίο ε, πολύ συγκεκριμένα θα λαμβάνει υπόψη και τον ιδιωτικό τομέα. Αυτές είναι ορισμένες από τις πτυχές του θέματος που θέλουμε να συζητήσουμε στην ομάδα υψηλού επίπεδου για τον τουρισμό. Από κοινού με τα κράτη-μέλη θέλουμε να διαπιστώσουμε όλοι ότι χρειαζόμαστε ένα στρατηγικό έγγραφο το οποίο όπως σας είπα θα συμπληρώσει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2010. Τον τουρισμό οφείλουμε να τον προσαρμόσουμε στην ψηφιακή κοινή αγορά. Ε, τέλη Μαΐου 2019 θα λάβει χώρα το Συμβούλιο Ανταγωνισμού και εκεί θέλουμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Στη Ρουμανία λοιπόν έχουμε προγραμματίσει τρεις ε, εκδηλώσεις και ελπίζουμε οι συζητήσεις αυτές ε, να ε, προάγουν ε, τα θέματα, τα συναφή με την προαγωγή του τουρισμού στα κράτη-μέλη. Ελπίζω όλοι από κοινού να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός διαφοροποιήθηκε ουσιαστικά όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Βιωσιμότητα λοιπόν είναι ένα καθοριστικό στοιχείο. στοιχείο που παίζει ρόλο στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα του περιβάλλοντος και της τεχνολογίας. Στη διάσκεψη για τον τουρισμό ε, που θα λάβει η χώρα αρχές Απριλίου στο Βουκουρέστι θέλουμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Στην Τούλτσα από τις 11 μέχρι τις 14 Ιουνίου θα έχουμε την Υπουργική Συνάντηση με θέμα στρατηγική για το Δούναμπι, στο Κεφρανιάντς στις 10 Απριλίου θα έχουμε μια συνάντηση του δικτύου Eden. Και στις τρεις αυτές εκδηλώσεις προφανώς και είστε προσκεκλημένοι. Ελπίζουμε μάλιστα να μπορέσετε να παρευρεθείτε. Η ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ορατή, αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε στην τεχνολογική εξέλιξη, η οποία και θα καθορίσει τον τουρισμό κατά τα επόμενα έτη. Προφανώς ε, και ε, από αυτές τις ε, τεχνολογικές δυνατότητες πρέπει να προσφέρουμε τουριστικές δυνατότητες. Ένα άλλο στοιχείο του τουρισμού είναι η ασφάλεια. Και για την ασφάλεια πρέπει να αγωνιστούμε όλοι από κοινού. Οι τουρίστες χρειάζονται πρώτα απ' όλα ασφάλεια. Και αυτό ε, αφορά την ε, ψυχαγωγία, αφορά την πολιτιστική περιέργεια και πολλά άλλα. Για το λόγο αυτό χρειαζόμαστε στρατηγικές σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, χρειαζόμαστε ένα σχέδιο για την ασφάλεια. Όλα αυτά βεβαίως αφορούν και τις τοπικές κοινότητες. Κοινωνική συνοχή. Αυτό είναι ένα καθοριστικό στοιχείο για τη Ρουμανία και όλα αυτά πρέπει να αντικατοπτρίζονται στα μέτρα τα οποία θα λάβουμε για τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω στο δεύτερο μέρος της ομιλίας μου να μίλησα λιγάκι πιο αργά. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ στους που κατάφεραν να σας παρακολουθήσουν. Ο κ. Λύρη, αντιπρόεδρο της ε, Task Force για το θέμα του τουρισμού. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, αγαπητέ Μπογκδάν, ευχαριστούμε πολύ. Λέω μιλτή στα ρουμανικά, είναι η μόνη λέξη που ξέρω στα ρουμανικά. Έχω πολλές ε, προσδοκίες από την Ρουμανική Προεδρία. Ελπίζω ότι το επόμενο εξάμεινο θα μιλήσουν στο Συμβούλιο πολύ περισσότερο για τουρισμό από τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό το λόγο προσκαλέσαμε και τον Υπουργό για να ανταλλάξουμε γνώμες. Αυτή η χρονιά θα είναι ιδιαίτερα σημαντική από πλευράς ε, της ευρωπαϊκής πολιτικής για τον τουρισμό και για τον τουρισμό γενικότερα. Ελπίζω η εργασία σας να είναι πολύ ορατές εντός του Συμβουλίου. Δηλαδή οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αντιληφθούν ότι πέραν οποιονδήποτε άλλων σημαντικών θεμάτων ή προτεραιοτήτων πρέπει να συζητείτε και το θέμα του τουρισμού. Εμείς οι ευρωβουλευτές είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε είτε επισήμως είτε ατύπως. Παρακαλώ πολύ ενημερώστε μας. Έχω μιλήσει επανειλημμένως με τον Υπουργό και έχουμε ενημερώσει όλες τις κυβερνήσεις ζητώντας τους να στηρίξουν την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο επιθυμούμε ένα κονδύλι ειδικά για τον τουρισμό. Η Ρουμανική Προεδρία πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτή η πρόταση θα προωθηθεί και ότι δεν θα διαμορφωθεί μια πλειοψηφική πρώτη, ε, θέση εναντίον της. Οπότε, παρακαλώ Υπουργέ, εστιάστε σε αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου μας. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί αυτό το ξεχωριστό κονδύλι από τον όχι επειδή είναι τεράστιο, αλλά για συμβολικούς λόγους. Το άλλο θέμα είναι το πώς η Ρουμανική Προεδρία εντός του Συμβουλίου θα μπορέσει να ενισχύσει το ρόλο του τουρισμού. Θα στηρίξω την Προεδρία και έχω μία ερώτηση. Στις 6 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι η... θα γίνει για πρώτη φορά η συνάντηση της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου. Υπάρχει δυνατότητα να συμμετάσχουμε και εμείς με κάποιο τρόπο. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, monsieur Ευχαριστώ πολύ. Α ακούσουμε μερικέ ερωτήσει και μετά α δώσουμε το λόγο στον Υπουργό. Κ. Βάντεν Κάμπ. Er, eh, ehm, Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχάς για τον ενθουσιασμό που δείξατε και την εξαιρετική σας παρουσίαση. Θα συμφωνήσω ότι εξαιτία ε, των ε, εξελίξεων και της μεγάλης σημασίας του τουρισμού στη βιομηχανία είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικαιροποιηθεί ο στρατηγικός ε, σχεδιασμός. Το έγγραφο από το 2010 χρειάζεται λοιπόν επικαιροποίηση και χαίρομαι πάρα πολύ ε, που αναφερθήκατε στο θέμα της υπερκάλυψης, ε, στο θέμα του υπερβολικού τουρισμού. Το ζούμε και στο Άμστερνταμ, τη Βαρκελόνη, το Λονδίνο. Αυτό είναι πραγματικά μεγάλο πρόβλημα όταν βλέπουμε ε, το πλήθος τουριστών με, τα διάφορα, με τις βαλίτσες τους, με τα Airbnb που κατακλείζουν τις πόλεις. Επίσης αναφερθήκατε στην ψηφιοποίηση αλλά και οι θεωρήσεις είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Όταν, ας πούμε, έχουμε 600 εκατομμύρια Κινέζους που θέλουν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη γιατί ανήκουν στη μεσαία τάξη και έχουν αυτή τη δυνατότητα, τότε μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει σε μια πόλη σαν το Βουκουρέστι. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε με τις θεωρήσεις σε αυτό το θέμα. Επίσης, μιλήσατε για την έλλειψη προσωπικού στην παρουσίασή σας και αυτό είναι το παράδοξο, κύριε Πρόεδρε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 500 εκατομμυρίων ε, κατοίκων δεν έχουμε αρκετούς ε, εργαζόμενους. Οι μισοί δεν είναι σε εργάσιμη ηλικία και οι υπόλοιποι πρέπει να ε, δουλεύουν και για τους άλλους. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε πως υπάρχει πρόβλημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις επαφές σας με τους ε, Φιλανδούς, με την επόμενη Προεδρία, είναι μία από τις προτεραιότητές σας, ακούσαμε, και ελπίζω να συνεχίσουν το δικό σας έργο τον Ιούλιο διότι έχουμε δει να επαναλαμβάνεται αυτό το λάθος, δηλαδή να κάνει δουλειά μια προεδρία και το επόμενο εξάμεινο η επόμενη να σταματά. Κυρία Μπιλμπάου, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Ευχαριστούμε που έτσι ενεργοποιήσατε ξανά το θέμα του τουρισμού. Ε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος εδώ σε αυτήν την Επιτροπή και είναι πολύ καλή ιδέα να επικαιροποιηθεί η ανακοίνωση της Κομισιόν του 2010, η οποία έχει λίγο απαρχαιωθεί. Επίσης με αρέσει που, μου αρέσει που θέλετε να δημιουργήσετε ένα φόρουμ μέσα στην ομάδα ανταγωνιστικότητας σε σχέση με την ανάπτυξη της απασχόλησης και την οικονομική δραστηριότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι, τα εργαλεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν ταιριάζουν σε εταιρείε που αναπτύσσονται, μικρές εταιρείε που αναπτύσσονται σε αγροτικές περιοχές εκτός των πόλεμων, σε περιοχές υπαίθρου. Τα εργαλεία που έχουμε μεταξύ αυτών και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία δεν ταιριάζουν σε αυτές τις επιχειρήσεις. Οπότε σωστή η κατεύθυνση προς την οποία κινείστε. Προφανώ δεν είναι αρκετό να γίνει αυτή η επικαιροποίηση αν δεν δοθεί συνέχεια μετά. Αναφέρατε όμως μερικά, μερικές προκλήσεις. Χρειάζεται μια εκστρατεία σε όλη την Ευρώπη. Όταν μιλάμε για βιωσιμότητα και συνοχή, θα πρέπει να σκεφτούμε ταυτόχρονα και το θέμα της μετανάστευσης και της προσαρμογής του όλου τομέα στα άτομα με αναπηρίες. Έχουμε 80 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιο είδου αναπηρία. Μια Ευρώπη που γυράσκει με το πέρασμα του χρόνου, οπότε χρειαζόμαστε καινούργια εργαλεία. Και θα ήθελα αυτά τα δύο θέματα, άτομα με αναπηρίες και μετανάστευση, να τα συμπεριλάβετε. Χρειαζόμαστε επίσης ανθρώπινο δυναμικό, καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό σε ένα τομέα το οποίο ζητάει εργατικό δυναμικό. Και μετά η ερημοποίηση. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες ερημοποιούνται, καταλείπονται, ενώ οι τουρίστες ψάχνουν όλο και περισσότερες φυσικές άθικτες περιοχές. Οπότε δεν θα πρέπει να παραμένουμε μόνο, να εστιάζουμε μόνο στις περιοχές που είναι πολιτική κληρονομιά. Άρα λοιπόν, μετανάστευση, άτομα με αναπηρίες και τρίτον, αυτό που σας είπα και το Brexit. Οι, τα Κανάρια νησιά έχουν το 25% των τουριστών που τα επισκέπτονται είναι από την ε, Βρετανία. Έχετε κάνει κάποια μελέτη, σκοπεύετε να κάνει κάποια μελέτη για ε, τις επιπτώσεις του Brexit στον τουρισμό και, και πώς θα επηρεάσει την απασχόληση και γενικότερα την οικονομία σε αυτές τις περιοχές. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Αμπιλμπάου. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κράμερ, θα πρέπει να σας αφήσω, διότι με περιμένουν σε άλλη συνεδρίαση. Θα ξανάλθω. Στο ενδιάμεσο θα με αντικαταστήσει ο κύριος Κορ, προσωρινά. Κύριε Κράμερ, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε για να μα παρουσιάσετε τι προτεραιότητε τη Προεδρία τονίσατε τη σημασία της βιωσιμότητας και της ποιότητας. Η βιωσιμότητα είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι ο, τουρισμό, ο υπερβολικός τουρισμός μπορεί να την καταστρέψει. Επίσης, Υπάρχουν και άλλοι τομείς του τουρισμού που αναπτύσσονται ταχύτατα τα τελευταία χρόνια. Ένας από αυτούς είναι και ο τουρισμός με ποδήλατο. Έχει αλλάξει τη μορφή του τουρισμού. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες αυξήθηκε κατά 20%. Είναι μια οικολογική μορφή τουρισμού που έχει και οικονομικές ε, επιπτώσεις. Υπάρχει μάλιστα μια μελέτη στην ε, Ελβετία που δείχνει ότι ο τουρισμός με ποδήλατο ε, δεν είναι μόνο ε, ίδιων των ε, φτωχότερων στρωμάτων, των φοιτητών κτλ. Ο ποδηλάτης κατά μέσο όρο δίνει περίπου 35 ευρώ την ημέρα πηγαίνοντας ε, στα δρομολόγια του. Επίσης, πάνω από... Οι, επίσης, οι διαδρομές με ποδήλατο, τα Velo Route έχουν αυξηθεί. Από 17 έχουν γίνει πάνω από 25. Για μένα η Σερβία αποτελεί υπόδειγμα σε ό,τι αφορά τις ε, διαδρομές με ποδήλατο στην περιοχή του Δούναβη. Υπάρχει εξαιρετική σηματοδότηση στις ε, διαδρομές 6 και 13. Οι πινακίδες είναι σε δύο γλώσσες, στα σέρβικα και στα αγγλικά και μάλιστα στα σύνορα υπάρχουν μεγάλες ε, πινακίδες που περιγράφουν τις ε, διαδρομές. Έχω κάνει ο ίδιος μου ποδήλατο την ίδια διαδρομή στην Ρουμανία και δεν βρήκα καμία τέτοια σηματοδότηση, ούτε προειδοποιητική σήμανση όταν πρόκειται να εισέλθει σε αυτοκινητόδρομο, ούτε τίποτα. Και η σε πινακίδες που ε, συνάντησα ήταν μόνο στη ρουμανική γλώσσα. Το πρόγραμμα αυτό είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ όμως δεν μπορούσα να διαβάσω τίποτα και να καταλάβω τίποτα. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο πολιτισμός και η ιστορία της ε, κάθε περιοχής από την οποία διέρχομαι. Οι Σέρβοι όμως ε, κατάλαβαν ότι ο τουρισμός με ποδήλατο μπορεί να αποφέρει έσοδα και έκαναν πράγματα γι' αυτό. Θεωρώ λοιπόν πως υπάρχει μέλλον και Μάλιστα η Σερβία μετά τις ε, προσπάθειες που έκανε για την ανάπτυξη του τουρισμού με ποδήλατο αύξησε τον αριθμό των τουριστών από, από 500 ε, σε 13.000 κάθε χρόνο και μάλιστα σε μία μέρα Ε, καθώς περνούσα από τη Ρουμανία, βγήκα ξαφνικά από τον ποδηλατόδρομο στον αυτοκινητόδρομο. Με προσπερνούσαν ταλίκες. Ε, από την άλλη μεριά ήταν οι ράγες του τρένου. Ήταν ε, φοβερά επικίνδυνη αυτή η κατάσταση. Ναι, μεν λοιπόν θέλουμε τον τουρισμό, την ανάπτυξη, όμως πρέπει να δώσουμε σημασία σε όλες τις μορφές, όπως και τον τουρισμό με ποδήλατο. Και θα ήθελα να σας κάνω μία πρόταση, μία σύσταση να καταβάλλετε προσπάθειες για να αυξηθεί η βιωσιμότητα του τουρισμού, όλες οι μορφές του τουρισμού και αυτό πιστεύω πως ε, θα δώσει ε, όθηση στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προσέξτε την εσήμανση θα πρέπει η σήμανση στο δρόμο, οι πινακίδε ε, να είναι Ε, Εντάξει, δεν είναι κατά ανάγκη υποχρεωτικό να είναι στη γλώσσα μου τα γερμανικά, αλλά μπορούν να είναι στα αγγλικά, σε μια γλώσσα που μπορούν να καταλάβουν περισσότεροι. Μιλώ για την ε, διαδρομή του Δούναβη στην ε, ρουμανική πλευρά. Η Ρουμανία έχει εξαιρετική και ε, εξαιρετικά αξιοθέατα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία της. Γι' αυτό λοιπόν θα ε, σας ε, παρότρινα να ε, κάνετε κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κράμερ. Το λόγο έχει κύριος Μαρινέσκου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Από την παρουσία σας ε, αυτό που αποκόμισα είναι ότι μέσα σε πέντε μήνες θα έχετε λύσει όλα τα προβλήματα. Όμως, έχω συγκεκριμένες ερωτήσεις για συγκεκριμένα ζητήματα. Τι πιστεύετε πως μπορούμε να καταφέρουμε ως προς ε, το έγγραφο αυτό στο Συμβούλιο ή στην ε, Κομισιόν. Αναφέρομαι στο επίσημο φυσικά έγγραφο με τη μορφή ανακοίνωσης ή ψηφίσματος αναφέρατε στην παρουσίασή σας ότι πρέπει και να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε στην πράξη αυτά που λέμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ρωτήσω τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρινέσκου. Η κυρία Τσαπαρντέλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα συζητούμε την ε, στήριξη του ευρωπαϊκού τουρισμού. Είναι ένα θέμα το οποίο ε, αγαπώ ιδιαίτερα. Ο κύριος Υπουργό είναι συμπατριώτης μου και προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ που θεωρούμε την ε, Ρουμανία μια χώρα με πολλές προοπτικές στον χώρο του τουρισμού. Και χαίρομαι επίση ε, για το ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ιδιαίτερα το Συμβούλιο, κατάλαβαν επιτέλου ότι ο τουρισμό χρειάζεται στήριξη. Στην Επιτροπή Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε δημιουργήσει μία task force, μία ομάδα λοιπόν για τον τουρισμό, στην οποία έχουμε συζητήσει αρκετές φορές την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ανάγκη για επικαιροποίηση αυτής. Όμως, δεν αρκεί μόνο η επικαιροποίηση. Η ανακοίνωση είναι από το 2010. Και τα τελευταία εννέα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συναντήσει νέες μόνο προκλήσεις στον τομέα του τουρισμού, αλλά και στην οικονομία και στην ε, Επιτροπή Τουρισμού εμείς αλλά και οι ε, διαφορές ε, ενώσεις θεωρούμε ότι αυτό που χρειάζεται είναι μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ευρώπη και η στρατηγική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους στόχους που συνδέονται με την ανάπτυξη του τουρισμού. Ταυτόχρονα χρειάζεται μια συγκεκριμένη ε, γραμμή χρηματοδότησης για τον ε, τουρισμό. Και αυτό ανεξάρτητα από την ε, διαφορά των απόψεων που επικρατούν. Πρέπει να συνδυαστεί αυτή η χρηματοδότηση και με την επικουρικότητα. Ο τουρισμός συνεισφέρει στο 11% του ΑΕΠ της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μην ξεχνάτε πως ε, έχουμε 1,2 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ε, τουρισμό. Γι' αυτό νομίζω πως δεν αρκεί μόνο να συζητούμε για την πολιτική επικουρικότητα, αλλά και να θέσουμε προτεραιότητες για την στήριξη του τουρισμού. Η Ρουμανία έχει, με την Προεδρία της έχει αναλάβει να ξαναφέρει το θέμα του τουρισμού στο Συμβούλιο και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ. Και νομίζω πως οι προσπάθειες αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα έγγραφο το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για, τις, ε, για το μέλλον του τουρισμού. Ελπίζω λοιπόν αυτό να μεταδοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και κάτι άλλο. Θεωρώ πως χρειάζεται κοινή πλατφόρμα για τη στήριξη του τουρισμού. Χρειάζεται μια κοινή λύση για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του υπερκερασμού ορισμένων πόλεων από τον τουρισμό. Υπάρχουν πάρα, πολλές, ε, πάρα πολλά μέρη στην Ευρώπη με μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον και νομίζω πόσο μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό και να αξιοποιηθούν τουριστικοί προορισμοί οι οποίοι είναι πολύ όμορφοι αλλά ελάχιστα γνωστοί. Γι' αυτό όμως χρειάζεται μία εξισορρόπηση στο, ε, στον ε, τουρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να στηρίξουμε ορισμένους τουριστικούς προορισμούς όπως ε, τα μοναστήρια του Μολδάβα, ε, το Δέλτα του Δούναβη, η διαδρομή των Καρπαθίων και άλλοι προορισμοί. Ελπίζουμε λοιπόν να αναπτυχθεί ο τουρισμός και άλλων περιοχών λιγότερο γνωστών. Επίσης υπάρχει και η πρόκληση της ψηφιοποίησης, η οποία ψηφιοποίηση αφορά και τον τουρισμό. Και θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό, αλλά και με την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων ε, όσων εργάζονται στον ε, κλάδο. Μπορούμε να κάνουμε διάφορες προσπάθειες μέσω διάφορων ε, προτάσεων, με πλατφόρμες που θα στηρίξουν ε, την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Σίγουρα έξι μήνες ε, δεν είναι αρκετοί, όμως ε, νομίζω πως μπορούμε να κάνουμε μια, ένα πρώτο βήμα για να αναπτύξουμε τον τουρισμό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ, Τίτερ. με, κύριε Υπουργέ. Εδώ είμαι πίσω για να με δείτε. Βέβαια η Κλάουδια, επειδή είναι από τη Ρουμανία, μίλησε για πολύ και με πολύ πάθο. Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι πιο σύντομη. Όσοι λοιπόν με γνωρίζουν από την Επιτροπή Μεταφορών, ξέρουν ότι ο Μίχαελ μιλάει πάντα για τα ποδήλατα και εγώ μιλάω πάντα για τα ποτάμια. Και αυτό θα κάνω και τώρα και ρωτώ πολύ συγκεκριμένα. Το βρίσκω πολύ καλό το ότι έχετε μια στρατηγική για την συνδιάσκεψη του, που θα έχει θέμα ο χώρο του Ντούναβη, ο ευρύτερο χώρο του Ντούναβη. Έχει ήδη οργανωθεί μια φορά, το έχει οργανώσει η Κλάουντια. Ο Δούναβη είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν γνωρίζω το κομμάτι του στη Ρουμανία. Και ερωτώ πολύ συγκεκριμένα όσον αφορά το υγροποιημένο φυσικό αέριο τα σκάφη, που με, τα πλοία που μεταφέρουν ε, υγροποιημένο φυσικό αέριο και διασχίζουν το Δούναβι. Ε, Πού ακριβώ βρίσκεστε, μήπω χρειάζεται κάποια βοήθεια χρηματοδοτική ενίσχυση από το εργαλείο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΕΦ. Επίση, όπω σα είπα, για τον δεν το ξέρω, έχετε και ένα κομμάτι τη μαύρη θάλασσα ε, που ε, αφορά τη Ρουμανία, ούτε αυτό το γνωρίζω. Ξέρω όμω ότι όλα αυτά μπορούν να πτυχθούν πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σα ρωτήσω, ε, τι είδου προβλήματα έχετε ενδεχομένω στο Ντούναβι και σε άλλε ακτέ με τη μόλυνση με πλαστικές ε, ουσίες, ε, γιατί αυτό το πρόβλημα το έχουμε εμείς, το χάρη, στη Γερμανία και νομίζω η μόλυνση με πλαστικά είναι κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να μπορέσουμε να ελέγξουμε. Ε, ευχαριστούμε την Γκεζίνα και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Μοντέρο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την παρουσία του εδώ στην Επιτροπή του Τουρισμού και βεβαίως ε, του εύχομαι στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχει στη διάθεσή του να μπορέσει να εφαρμόσει αυτό το αρκετά φιλόδοξο πρόγραμμα που μας ε, παρουσίασε. Ε, διαπίστωσα με ικανοποίηση ότι αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η Ρουμανική Προεδρία θα αντιμετωπίσει τον τουρισμό ως προτεραιότητα. Θα συμπεριλάβει και την ανταγωνιστικότητα. Άρα δηλαδή αναγνωρίζουν ότι ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός ε, για την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά διάρκεια των πέντε ετών, όπως ε, θα ακούσατε, υπάρχουν εδώ συνάδελφοι οι οποίοι δούλεψαν πολύ σκληρά έτσι ώστε ο τουρισμός να μπει στην πρώτη βαθμίδα της ευρωπαϊκής ε, κλίμακας. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι είναι σημαντικό και εσείς ε, κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας σας να προβάλλετε τον τουρισμό ως καθοριστική σημασία για την οικονομία, για τις περιοχές μας και για την Ευρώπη. Κατόπιν, όσον αφορά στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, παρουσίασε τη χρηματοδότηση για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. 330 εκατομμύρια ευρώ και τώρα το Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει το ποια θα είναι η δική μας η γραμμή για τους ε, συγκεκριμένους ε, παίκτες. Είναι λοιπόν ανόητο και δεν έχει κανένα νόημα να αναφέρουμε συγκεκριμένες προκλήσεις. Και θα πρέπει να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα για αυτές τις προκλήσεις. Εγώ θέλω να αναφερθώ στην ψηφιοποίηση και στο Brexit. Καταρχήν ψηφιοποίηση βρισκόμαστε, ζούμε μια πραγματική ψηφιακή επανάσταση. Οπότε η ψηφιοποίηση θα πρέπει να τεθεί στην υπηρεσία των πολιτών μας. Αν σκεφτούμε ότι ο τουρισμός δημιουργεί τεράστιο αριθμό θέσεων εργασία, αν η ψηφιοποίηση τεθεί στην υπηρεσία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 20% αυτών συνδέονται με τον τουρισμό στην Ευρώπη, καταλαβαίνετε ότι θα είναι τρομακτικό το όφελος. Χρειαζόμαστε όμως εργαλεία στο πλαίσιο προγραμμάτων που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουρισμού και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Έχουμε μία καινούργια γενιά η οποία ήδη έχει προσόντα ή αυτή τη στιγμή αποκτά προσόντα σε σχέση με την ψηφιοποίηση και πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η νέα γενιά για να καλυφθούν κενά που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στον τομέα του τουρισμού στην ψηφιοποίηση. Μόνο έτσι θα αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρησιών μας. Ο δρόμος είναι μακρύς. Επίσης, ε, σε σχέση με τους προορισμούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή δέχονται υπερβολικά μεγάλους αριθμούς τουριστών. Είναι θέμα διαχείρισης. Τα 27 κράτη-μέλη θα πρέπει να ενημερωθούν ενδεχομένως με μια επιστολή έτσι ώστε όλα αυτά που λέμε σήμερα εδώ να τα γνωρίζουν. Να κάνουμε από κοινού μια προσπάθεια για μια Ευρώπη πιο ευφύ, πιο έξυπνη, με έξυπνε ευφύ πόλεις, ευφύ προορισμούς και μια καλύτερη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την ε, κυρία Μοντέρο. Ε, στο τέλος ε, αναφέρομαι εγώ στον κατάλογο. Εγώ θα δείξω πολύ σύντομα δύο θέματα τα οποία η πολιτική μας ομάδα έχει αναφέρει για τα σύνορα. Καταρχήν τα δικαιώματα των επιβατών στις αέριες μεταφορές. Αυτό το θέμα υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό στο Συμβούλιο. Θέλουμε να ξέρουμε τι θα κάνετε εσείς. Δεύτερον, έχουμε μιλήσει για το τις πολυλειτουργικές, πολυτροπικές μάλλον μεταφορές, δηλαδή να έχει κανείς ένα εισιτήριο από το σπίτι του, να μπορεί να πάει ε, μέχρι, με το ταξί μέχρι το αεροδρόμιο, να χρησιμοποιεί άλλα μέσα και θέλω να ρωτήσω, όσον αφορά αυτή τη δυνατότητα ταξιδιού, έχετε σημειώσει εσείς κάποια πρόοδο. Αυτά είχα να ρωτήσω. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, φαντάζομαι τελειώστε με τι ε, σημειώσει σα και παρακαλώ έχετε το λόγο για να απαντήσετε σε όλε αυτέ τι πολλέ ερωτήσει που ετέθησαν. Ε, Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Είναι πολύ ποιοτικέ ερωτήσεις. Θα τις απαντήσω μία προς μία. Σας καλώ σε τρία σε τρεις εκδηλώσεις που ε, θα διοργανώσουμε στη Ρουμανία οπότε θα μάθετε και περισσότερα ρουμανικά λέω στον κύριο συνάδελφό σας ο οποίος ε, <laughs> είπε ότι ε, ξέρει μόνο μία ρουμανική λέξη και έτσι κι αλλιώς τον ευχαριστώ βέβαια αλλά μπορεί να μάθει περισσότερες η Ρουμανία είναι μια πολύ όμορφη χώρα δεν θέλω να <laughs> τη διαφημίσω βέβαια αλλά έτσι κι αλλιώς μεροληπτικός είμαι, αλλά έχουμε εξαιρετικά βουνά, μεγάλη βιοποικιλότητα, πολύ πλούσια. Τα Καρπάθια, το Δέλτα του Δούναβη είναι περιοχές ε, πολύ μεγάλου φυσικού κάλους. Πύργους, κάστρα, μοναστήρια, εκκλησίες που είναι πολιστική κληρονομιά της UNESCO να μας επισκεφτείτε. Θα μείνετε εντυπωσιασμένοι. Τώρα, το θέμα της χρηματοδότησης του τουρισμού, της επαρκούς χρηματοδότησης του τουρισμού. Τα 300 εκατομμύρια ευρώ που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, είναι μια σημαντική η απόφαση θα ληφθεί από τους ε, αρχηγού κρατών κυβερνήσεων. Αυτοί θα αποφασίσουν να θα δημιουργηθεί μια γραμμή στον προπολογισμό για τον τουρισμό. Οπότε ξεπερνάει τις συζητήσεις του Συμβουλίου Υπουργών ε, Ανταγωνιστικότητας. Χρειαζόμαστε Επίσης ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τον βιώσιμο τουρισμό. Η Κομισιόν ακόμα δεν έχει λάβει τέτοια, αναλάβει τέτοια πρωτοβουλία. Πρέπει ο τουρισμός να είναι πιο ορατός επιτέλους στην ημερήσια διατάξη της Ευρώπης. Είναι πολύ σημαντικός για την οικονομία μας. Οπότε για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια θα προτείνουμε συμπεράσματα του Συμβουλίου για τον τουρισμό, ειδικά ιδιαίτερα συμπεράσματα εντός του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας. ο τουρισμός χρειάζεται οικονομική στήριξη και ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο. Θέλουμε λοιπόν να στηρίξουμε οικονομικά τον τομέα. Εκεί συμφωνούμε μαζί σας λοιπόν πλήρως. Μετά, Το θέμα των θεωρήσεων. Είναι θέμα που αφορά και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ασφαλώς και θέλουμε μεγάλους αριθμούς, ε, μεγάλο αριθμό τουριστών στην Ευρώπη. Περιμένουμε τα συμπεράσματα της αρμόδιας επιτροπής πρώτα και μετά θα δούμε το θέμα πολύ σοβαρά. Θα λάβουμε υπόψη τα συμπεράσματα της αρμόδιας επιτροπής να δούμε ποιες είναι, ποια είναι τα πλεονεκτήματα για τον τουρισμό ε, και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε και την ευρωπαϊκή κουλτούρα. Μετά, η κυρία Μπιλμπάου. Χαίρομαι που μιλήσατε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειάζεται να έχουμε μια κοινή πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να τις στηρίξουμε. Σε ό,τι αφορά τα 80 εκατομμύρια ατόμων που έχουν κάποια αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει σίγουρα να σκεφτούμε το πρόβλημά τους και ενδεχομένως να τους δώσουμε και την ευκαιρία να εργαστούν στον τουριστικό τομέα. Κύριε Κράμερ, Μιλήσατε για το βιώσιμο τουρισμό. Ασφαλώς και θα πρέπει η ιδέα της βιωσιμότητας να είναι κεντρική στη σκέψη μας. Αυτή τη στιγμή η βιωσιμότητα αφορά μόνο τις προστατευόμενες φυσικές περιοχές. Για παράδειγμα, Natura 2000. Δεν θα πρέπει όμως να περιοριστούμε εκεί. Η βιωσιμότητα θα πρέπει να ενταχθεί στο σχέδιά μας για όλες τις τουριστικές περιοχές. Μετά, οι ποδηλατόδρομοι και ο τουρισμός ποδηλάτου. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα. το ποδήλατο είναι άσκηση και ταυτόχρονα προστατεύει το περιβάλλον. Δώσατε ένα παράδειγμα λίγο αρνητικό για τη Ρουμανία. Έχετε δίκιο. Η Ρουμανία δεν είναι ακόμα έτοιμη. Δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα πλήρως στις απαιτήσει του ποδηλατικού τουρισμού. Παρ' όλα αυτά σιγά σιγά γίνεται προτεραιότητά μας. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε τα νομοθετικά κείμενα που χρειάζονται προκειμένου να οριστούν, ή να καθοριστούν ποδηλατικές διαδρομές που θα επιτρέπουν στον τουρίστα να μην αναμειγνύεται, στον ποδηλάτη να μην αναμειγνύεται με αυτοκίνητα. Προσπαθούμε να εντάξουμε τη Ρουμανία στις ευρωπαϊκές ε, διαδρομ, ποδηλατικές διαδρομές. Ευχαριστώ πολύ για την όμορφη περιγραφή που κάνατε για τα τοπία της Ρουμανίας, για το τουριστικό της προϊόν. Και ελπίζω ότι θα σας ξαναβρούμε στη Ρουμανία σε μια ποδηλατική διαδρομή, σε ένα ποδηλατόδρομο και θα μπορέσετε να επισκεφθείτε καλύτερα τη χώρα μου. Κύριε Μαρινέσκου. Με ρωτήσατε τι θα κάνουμε στην πράξη. Προφανώς δεν είναι δική μου η απόφαση. Εγώ θα ήθελα να δούμε απτό αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια του εξάμεινου της Προεδρίας μας. Σίγουρα θα συζητήσουμε πολλά θέματα, θα εντοπίσουμε λύσεις. Πρέπει όμως να συμφωνήσουμε όλοι. Και παρακαλώ πολύ εμπιστευτείτε μας. Είστε Ρουμάνος, αγαπάτε τη Ρουμανία, οπότε να είστε σίγουροι ότι η Ρουμανική Προεδρία θα φέρει θετικά αποτελέσματα για τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Έτσι ώστε η Ευρώπη να παραμείνει ο υπαριθμόν ένα τουριστικός προορισμός στον κόσμο. Κυρία Ταπαρδέλ, στρατηγική μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χαίρομαι που μιλάμε την ίδια γλώσσα. Χρειαζόμαστε μια ενιαία προσέγγιση για τον τουρισμό στην Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και αδύνατο. Θα εξετάσουμε τη δυνατότητα το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα να επεξεργαστεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τον τουρισμό. Θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η στρατηγική του 2010 διότι έχουν γίνει τόσες πολλές αλλαγές, ε, έχει προχωρήσει τόσο πολύ ο κόσμος ε, τα τελευταία 20 χρόνια που χρειάζεται επικαιροποίηση. Το θέμα των πλωτών οδών. Είναι αλήθεια ότι ο Δούναβης είναι εξαιρετικός προορισμός για τους τουρίστες. Και μάλιστα το πιο εντυπωσιακό κομμάτι του Δούναβη είναι αυτό της Ρουμανίας, σας βεβαιώ. Οι υποδομές μας δεν είναι άριστες βέβαια, αλλά θα οργανώσουμε μία διάσκεψη για τον Δούναβη. Θα έχετε την ευκαιρία να έρθετε και να δείτε πόσο όμορφος είναι πραγματικά ο Δούναβης. Ε, είναι ένα σημείο, ένα μέρος το οποίο είναι πολύ κληρονομιά της UNESCO. Παραδοσιακό μέρος. σε αυτή τη διάσκεψη θα συζητήσουμε το πώς θα γίνει πιο ελκυστικός ο ποτάμιος τουρισμός. Τέλος, Προς την κυρία Μοντέρο νομίζω, απαντώ. Η ανάπτυξη του τουρισμού, η συμβολή του τουρισμού στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Ο τουρισμός είναι ένας από τους κλάδους που πιο πολύ συνεισφέρουν στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ. Πάνω από 10% του ΑΕΠ. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε φτάσει στο, στη μέγιστη δυνατότητά μας. Στην ομάδα ανταγωνιστικότητας θα θέσουμε αυτό το θέμα έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε όλες μας τις δυνατότητες, το 100% του δυναμικού μας. Και μου απομένει μια ακόμα ερώτηση. Ε, τις συνδυασμένες μεταφορές είναι μια πολύ καλή ιδέα, θα διευκόλυνε πολύ τους τουρίστες. Ευχαριστώ για αυτή την ιδέα, δεν την είχαμε σκεφτεί. Θα την εξετάσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Ε, και μην ξεχνάτε και τα δικαιώματα των επιβατών στις ενέργειε μεταφορές, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που είπατε, για τις απαντήσεις που δώσατε στις ε, ερωτήσεις. Ε, σας συγχαίρω γιατί πραγματικά παρουσιάσατε με ιδιαίτερη επιτυχία το τι κάνει η χώρα σας στον τομέα του τουρισμού. Καλή επιτυχία γιατί η δική σας επιτυχία είναι και δική μας.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 Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Αφήνουμε λιγάκι την Προεδρία, τη Ρουμανική και περνάμε σε ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ του πολίτε ε, και βλέπω ότι αρχίζουν και έρχονται όλο και περισσότεροι συνάδελφοι γιατί ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Ε, πρόκειται για την κατάργηση κάθε χρόνο τη χειμερινή και τη θερινή ώρα. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, στην κυρία Σκοκ, για να μα παρουσιάσει την έκθεσή τη. Παρακαλώ. Thank you, Chair. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω ολοκληρώσει το σχέδιο έκθεσης για την εποχιακή αλλαγή ώρας. Το Δεκέμβριο το ολοκλήρωσα. Με συγχωρείτε, αλλά αν θέλετε να αποχωρήσετε από την αίθουσα, παρακαλώ γρήγορα και ήσυχα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχω ολοκληρώσει λοιπόν το σχέδιο έκθεσης για την εποχιακή αλλαγή ώρας, ήδη το Δεκέμβριο. Παρουσιάστηκε εδώ τον Ιανουάριο στην Επιτροπή και δέχτηκα τη στήριξη πολλών μελών Έκτοτε έχουμε λάβει 76 τροπολογίες από σχεδόν όλες τις πολιτικές ομάδες και χαίρομαι πολύ που βλέπω μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Η εποχιακή, η πρόταση για την ε, αλλαγή προκύπτει από πρωτοβουλία των πολιτών και κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης ε, είχαμε πληθώρα από αντίσεων και μεγάλη ανταπόκριση από τους πολίτες. Έγιναν διμερείς ε, συναντήσεις με τους ε, σκιώδεις εισηγητές, μία άτυπη συνάντηση και χθε μία τακτική. Χθε παρουσιάστηκαν οι διαφορετικέ επιλογές για του και εισηγητέ, έτσι ώστε να γίνουν δεκτέ οι περισσότερε τροπολογίες. Και βλέπω με μεγάλη μου χαρά ότι η χθεσινή συνεδρίαση πήγε πολύ καλά. Είχαμε την ε, πλήρη στήριξη όλων των σχεδόν εισηγητών για τους ε, συμβιβασμούς τους οποίους καταλήξαμε. Θα στηρίξουμε λοιπόν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το σχέδιο έκθεσης στο οποίο είμαι εισηγήτρια ε, αναφέρεται σε αυτό, στην ε, κατάργηση της αλλαγής εποχιακής ώρας. Χρειάζεται όμως να επιλέξει το κάθε κράτος μέλος, μια που είναι εθνική αρμοδιότητα, την ε, ώρα την οποία θα ακολουθήσει και θα πρέπει να συσταθεί ένας συντονιστικός μηχανισμός, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη μεταξύ τους να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για μια εναρμόνιση έτσι ώστε η εσωτερική αγορά, οι μεταφορές και οι τηλεποκοινωνίες να είναι εναρμονισμένες. Καθώς επίσης και να προβλεφθεί μία μεγαλύτερη περίοδος προσαρμογής. Κάτι που δεν έτυχε τη στήριξη όλων είναι το πότε θα καταργηθεί η εποχιακή αλλαγή ώρα. Εγώ θα προτιμούσα αυτό να γίνει το 2021, έτσι ώστε όλα τα κράτη-μέλη και οι αρμόδιοι να προετοιμαστούν καταλήλως για να οργανωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ενιαία αγορά και να αποφύγουμε τις αρνητικές επιπτώσεις για τους πολίτες. Ωστόσο, οι χθεσινές ε, συζητήσεις έγιναν χωρίς τις άλλες έξι επιτροπές που θα γνωμοδοτήσουν στην έκθεση αυτή, οι οποίες θα ψηφίσουν αυτή τη βδομάδα. Γι' αυτό το λόγο την επόμενη εβδομάδα θα γίνει άλλη μια συνάντηση των σκιωδών εισηγητών, ώστε να συζητήσουμε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στις άλλες έξι επιτροπές. Νομίζω πως μπορούμε να συνεχίσουμε και να τηρήσουμε το προτινόμενο χρονοδιάγραμμα, έτσι ώστε να ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή στις 4 Μαρτίου. Είναι σημαντικό να γίνει αυτό, διότι πρέπει το Κοινοβούλιο να καταλήξει σε μια απόφαση πριν τις εκλογές, αλλά και να παρουσιάσει τα, εργα... τα αποτελέσματα των εργασιών του μέχρι τότε. Ελπίζω λοιπόν να συνεχιστεί η καλή συνεργασία που είχαμε με τους υπόλοιπους κοιόδες εισηγητές και κλείνοντας θα πω ότι είμαι αισιόδοξη ω προς το χρονοδιάγραμμα και ως προς την ε, ευκαιρία που θα έχουμε να προσφέρουμε έργο στους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ουλσκοκ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές. Πρώτα έχει το λόγο το ΕΛΚ και ο κύριος Σβόμποντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς την εισηγήτρια, κυρία Ούλσκογκ, για τη δουλειά που έκανε και πράγματι στη χθεσινή συνάντηση των σχεδόν εισηγητών καταλήξαμε σε ένα σαφές αποτέλεσμα. Αυτά δηλαδή που σας ε, παρουσίασε μόλις η εισηγήτρια. Να προσθέσω επίσης ε, σε αυτά που είπε η κυρία Ουλφσκόγκ ότι η θέση στην οποία καταλήξαμε δεν ήταν αποτέλεσμα πρωτοβουλίας πολιτών, ήταν μια επιτυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διότι χάρη στην δική μας δουλειά και, την, ε, και τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε, από το μηδέν φτάσαμε στην νομοθετική διαδικασία. Η κυρία Ούλσκο ανέφερε ότι υπάρχουν άλλες έξι επιτροπές που θα γνωμοδοτήσουν και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων η ψηφοφορία χθες ήταν ε, πολύ θετική. Αυτά ε, ως ε, πρόεδρος της Επιτροπής Γιούρη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σβόποντα. Θα δώσω το λόγο στους ECR. Ε, Ο κύριος Λωτόφσκι λείπει, αλλά έχει ορίσει την καταστάτη. Ναι, γεια σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα διαβάσω το κείμενο του σκιώδου εισηγητή. Καταρχάς, ε, ο κ. Ζωτόφσκι ευχαριστεί πάρα πολύ. Η ομάδα ECR θεωρεί πως η πρόταση να καταργηθεί η εποχιακή αλλαγή ώρας είναι αρκετά καλή. Οι συμβαστικές ε, τροπολογίες επίσης. Η ομάδα ECR θεωρεί ότι οποιασδήποτε αλλαγές ε, στην εποχιακή ώρα θα πρέπει να συνοδευτούν από εκτίμηση αντικτύπου και ειδική ομάδα. Επίσης, συμφωνούμε με την άποψη της εισηγήτριας ότι χρειάζεται μία επικοδομητική προσέγγιση για να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές καθώς και συντονισμός έτσι ώστε να ε, διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της ε, νέας αγοράς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπιλμπάου εκ μέρους των Φιλελευθέρων. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ επικοδομητική δουλειά που έχει κάνει και την συνεργασία με όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Είναι καλό μέτρο η αναβολή του μέτρου της κατάργησης μέχρι το 2021 γιατί πράγματι τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση Μερικές χώρε ήδη έχουν δημιουργήσει ομάδες εργασία που αναλύουν ε, από πολλές ε, οπτικές γωνίες τις επιπτώσεις. Γι' αυτό και εμεί ζητούσαμε την αναβολή μέχρι το 2021. Το έχουμε πει στο παρελθόν και το επαναλαμβάνουμε. Αυτός ο μηχανισμός συντονισμού θα πρέπει να λειτουργεί σωστά. θα μας επιτρέψει να κάνουμε μία ανάλυση όλοι μαζί και η Κομισιόν θα πρέπει να παίξει συντονιστικό ρόλο. Θα πρέπει να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα του ποια αλλαγή της ώρας θα καταρριθεί. Η του φθινοπόρου ή της άνοιξης, του χειμώνα ή του καλοκαιριού, έτσι ώστε να είμαστε συνεπείς μεταξύ μας. Θα επαναλάβω αυτό που είπα παλιότερα. Η ημερίδα που οργανώσαμε ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Αναλύσαμε ε, θέματα που έχουν σχέση με την ενέργεια, για παράδειγμα. Και, ο, και η η ανέφερε ότι παλιότερα έχει αποφασιστεί η εποχιακή αλλαγή για ενεργειακούς λόγους. Αυτή τη στιγμή όμως δεν γίνεται κανενός είδους ε, εξοικονόμηση ενέργειας. Θέματα τα οποία προκύπτουν δευτερευόντως όπως αυτό των μεταφορών μπορούν να λυθούν εύκολα. Οπότε είναι προφανές ότι οι βλάβες που προκαλούνται στην υγεία είναι πιο σημαντικές από τα ωφέλη που προκύπτουν. Και όλο και πιο σημαντικές. Η λαϊκή πρωτοβουλία στην οποία συμμετείχαν πάνω από 4,6 εκατομμύρια άτομα ήταν πάρα πολύ σημαντική, οπότε θα πρέπει να δώσουμε μια συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μπιλμπάου, σας ευχαριστώ πολύ και για την αισιοδοξία σας. Κύριο Στέρντ έχει το λόγο από τους ε, Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς την εισηγήτρια για τις δύο επιλογές που μας έδωσε σχετικά με τις συμβαστικές τροπολογίες. Η πράσινη είναι ευχαριστημένη διότι φαίνεται πως υπάρχει μια ευρεία συνένεση για την πρώτη επιλογή. Το θέμα είναι να γίνει συζήτηση για το πώς πρέπει να γίνει η εναρμόνιση της διακοπής αλλαγής εποχιακής ώρας και για να μην καταλήξουμε σε μια κατακαιρματισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τις ε, ζώνες Χρειάζεται λοιπόν να διασφαλιστεί η συνέχεια και η ομαλή λειτουργία της ε, ενιαίας αγοράς, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι μεταφορές ε, και η δημόσια υγεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να καθυστερήσει την εφαρμογή της ε, κατάργησης της εποχικής αλληλής ώρας εφόσον διαπιστώσει ότι τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Τώρα, για το αν θα διατηρηθεί η θερινή ή χειμερινή ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συστήσει μια ομάδα πυρογνωμόνων που θα καταλήξει σε προτάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ταλούντε Για του, την ομάδα EFDD, κυρία Γιούτο, θέλετε να πείτε κάτι ή συζητάτε ακόμα. Κυρία Αγιούτο, όχι, δεν θέλετε να μιλήσετε. Ωραία, κυρία Μάισνερ ε, έχει το λόγο, εφόσον η κυρία Γιώτο δεν θέλει να τοποθετηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την ε, εισηγήτρια και τους κοιόδης εισηγητές για την καλή δουλειά τους. Θεωρώ πως το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, όχι μόνο στη δική μας επιτροπή, αλλά και σε άλλες επιτροπές. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί που θεωρούν ανοησία αυτό το θέμα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, βέβαια, από όσο είμαι ευρωβουλευτής και εγώ προσπαθώ να πιέσω για την κατάργηση της εποχιακής αλλαγής ώρας. Έχω μιλήσει και με την κυρία Μπούλτ για τον ε, φόβο που υπάρχει πως θα προκύψουν θα προκύψει κατακαιρματισμό στην Ευρώπη λόγω των, της διαφορετικής ώρας που θα ακολουθεί κάθε χώρα. Χρειάζεται όμως να διερευνήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε για να επιλέξει το κάθε κράτος μέλος την ε, ώρα που θέλει. Τώρα, ως προς το θερινή ή ε, χειμερινή ώρα, στην ε, Ελβετία έγινε ένα δημοψήφισμα και η, πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε να μην αλλάξει τίποτα. Το θέμα βέβαια είναι να έρθουμε λίγο στα λογικά μας, ε, διότι η Ρωσία και η Κίνα έχουν ήδη καταργήσει τις εποχιακές αλλαγές ώρες διότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι, ιατρικοί λόγοι, οι βιολόγοι έχουν διαπιστώσει επιστημονικά ότι δεν είναι καλό για την ανθρώπινη υγεία να αλλάζει η ώρα δύο φορές το χρόνο. Και νομίζω πως υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι εκτός από αυτό για τις ε, μεταφορές, για παράδειγμα, ε, για ε, τους ε, μαθητές που πηγαίνουν στο σχολείο. Υπάρχουν άπειροι λόγοι λοιπόν να καταργηθεί η εποχιακή αλλαγή ώρας ε, και ε, νομίζω πως ε, δεν θα οδηγηθούμε πουθενά αν προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε με τα κρατη αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα σωστό, καλό αποτέλεσμα και ένα σαφή προσανατολισμό πριν λήξει αυτή η κοινοβουλευτική θητεία έτσι ώστε να ε, βοηθήσουμε όσους υποφέρουν από αυτές τις εποχιακές αλλαγές της ώρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ρικέ, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής. με την πίεση της ε, πρωτοβουλίας αυτής των πολιτών τίθεται το ερώτημα αν θα συνεχίσουμε με τις αλλαγές, ε, τις εποχιακές αλλαγές η πλειοψηφία λέει ότι θα είναι καλύτερο να σταματήσουμε αλλά υπάρχει και αντίθετη γνώμη δεύτερον πού θα σταματήσουμε, ποια θα καταργήσουμε την χειμερινή ή την ε, θερινή αλλαγή και τρίτον και, και αυτό δεν είναι πολύ σοβαρό το σοβαρό είναι το τρίτο, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αρμοδιότητα για το θέμα αυτό. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιβάλλει μια εναρμόνιση. Μπορούμε να αναμένουμε ότι κάθε κράτος μέλος θα αποφασίσει από μόνο του για την ώρα του. Σε συνάρτηση και με το που ακριβώς βρίσκεται γεωγραφικά. Οπότε μπορεί να δημιουργηθεί ένα μικρό χάος, μια σύγχυση. Αυτό μπορεί να έχει επιπτώσει στις μεταφορές των προσώπων, των αγαθών, εμπορευμάτων κλπ. Οπότε, ε, για τις δύο πρώτες ερωτήσεις υπάρχει αφορά απόψεων, αλλά για την τρίτη, ότι χρειάζεται, πολύ, ε, ότι χρειάζεται εναρμόνιση, Όλοι συμφωνούμε. Δημιουργήθηκε έτσι ένας πυρετός και ένας φοβερός ενθουσιασμός ότι πρέπει να βιαστούμε κλπ. Αλλά αυτή η βιάση μπορεί να μας οδηγήσει σε ε, σύγχυση. Οπότε θα ήθελα να ψηφίσουμε κατά της πρότασης αυτής. Η Κομισιόν έχει κάνει μελέτες αντικτύπου. Θα μπορούσε να μας ενημερώσει τι περιμένει ως εναρμόνιση από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Ντομινίκ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον ε, κύριο Βαντάλ. Πίτερ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, Στην ε, Ολλανδία πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να υποπέσουμε σε λάθη. Ε, φοβάμαι ότι στην Ευρώπη θα προκύψει μια εμβαλωματική κατάσταση. Οι μεν θα κάνουν το Α, οι άλλοι το Β. Η Κομισιόν επί του θέματο δεν έχει αρμοδιότητα. Με άλλα λόγια, περνάμε από τη σκύλα στη χάριβδη. Και γι' αυτό λοιπόν εγώ το λόγο προτείνω να μην κάνουμε τίποτα γιατί δεν ξέρουμε καν ποιες θα είναι οι συνέπειε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμα σωστή ανάλυση, εμβριθής ανάλυση. Στην Ευρώπη τι προτείνουμε, σας είπα, εμβαλωματική λύση, συμβιβασμούς, μετά σκεπτόμαστε κάποιο μηχανισμό, μετά λέμε η Κομισιόν αποφασίσει, η Κομισιόν όμως δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα. Κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι υπέρ της τροπολογίας υπαριθμών 19 των συναδέλφων Ρίλ και Κεβαντάλ μεταξύ άλλων. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, πρέπει να απορριφθεί. Καλύτερα λοιπόν να διορθώσουμε έστω τα μισά από το να κάνουμε σοβαρά λάθη. Ευχαριστούμε. Πίτα, ο Βιμ είναι ο επόμενος. Αυτά που είπε το ρητό υποτίθεται από την Ολλανδία, το έχεις ακούσει ποτέ. Κύριε Βιμ, ε, κοιτάξτε, το ρητό αυτό δεν είναι από την Ολλανδία, αλλά είναι από τις κάτω χώρες. Άλλο η Ολλανδία, πρόεδρε, άλλο οι κάτω χώρες. Εγώ δεν είμαι από την Ολλανδία, είμαι από τις κάτω χώρες. Λοιπόν, Πρόεδρε, έχω μόνο μία ερώτηση προς τον εισηγητή. Πότε πρόκειται να ολοκληρωθεί αυτό το θέμα. Γιατί για να είμαι ειλικρινής, ο κύριος Βαντάλεν είπε αυτά που είχα και εγώ κατά νου. Τώρα, τι γίνεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και τρία χρόνια συζητά για το θέμα αυτό. Ο κύριος Γιούνκα μας ε, έδωσε μία χοντρή πατάτα που δεν είναι καν μαγειρεμένη. Ένα κομμάτι κρέας αν θέλετε που δεν το έχουμε μαγειρέψει. Αν λοιπόν μιλάμε και εφόσον μιλάμε ε, για την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι είναι ντροπή το ότι έχουν περάσει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια πριν να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Αυτή λοιπόν είναι η μόνη ερώτηση που έχω να κάνω προς τον εισηγητή. Πέστε μας, πότε πρόκειται επιτέλου να ολοκληρωθεί το θέμα αυτό και με κάποιο αποτελεσματικό και σωστό τρόπο. Ευχαριστούμε και για τα εισαγωγικά, τα διευκρινιστικά που είπες. Ο κύριος Κράμα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Πολλοί φοβούνται αυτό το μοσαϊκό, την εμβαλωματική λύση που αναφέρθηκε προηγουμένως στην Ευρώπη και πολλοί προσποιούνται ότι δεν ισχύει αυτό. Μα συγγνώμη, τρεις ε, ζώνες ορών έχουμε στην Ευρώπη και εγώ διαρωτώ με πώς γίνεται να υπάρχει διαφορετική ώρα ανάμεσα στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Αυτό είναι τελείως τρελό. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με γεωγραφική τοποθέτηση. Εγώ σας το λέω ως Γερμανός. Όταν οι Γερμανοί κατήχαν, ε, έβαλαν σε κατοχή τη Γαλλία, αποφάσισαν κοινή ώρα. Και μετά ο Χίτλερ με το Φράνκο ε, συνήψαν συμφωνία και είπαν ίδια ώρα και στην Ισπανία. Γι' αυτό λοιπόν αυτές οι χώρες είναι στην ίδια ζώνη ώρα και έχουμε του δυτικού. Ιρλανδία, Πορτογαλία, ε, Μεγάλη Βρετανία, άρα δηλαδή άλλη ώρα. Από την άλλη έχουμε την Ελλάδα που πάει στην ίδια ώρα με τις χώρες της Βαλτικής, αλλά όχι με τις βόρειες γειτονικέ της χώρας, παρότι η Ελλάδα θα έπρεπε κανονικά να πάει σε άλλη ζώνη ώρας. Άρα δηλαδή το πρόβλημα υφίσταται, είναι ένα μοσαϊκό, μια εμβαλωματική λύση, ενδέχεται να μην αποκτήσουμε μία ζώνη για την Ευρώπη, αλλά ακόμα και εάν δεν επιτύχουμε τίποτα, το να συνεχίσουμε να εξετάζουμε τι συμβαίνει είναι σημαντικό. Ε, δεν θέλουμε αυτή την εμβαλωματική λύση. Υπάρχει ε, ένα patchwork και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά το να σταματήσει πια το να αλλάζουμε την ώρα. Επιτέλους αυτό πρέπει να το πετύχουμε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κράμα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο κύριος Ρικέ. Δηλαδή αυτά που είπε σχετικά με το πώς μπορεί να πετύχει όλη αυτή η διαδικασία εναρμόνισης. Διότι η συγγήτρια είπε ότι υπάρχει ένας ε, συντονισμός, ένας μηχανισμός συντονισμού ο οποίος προβλέπεται, το είπε η κυρία Ουλσκοφ. Αλλά λαμβάνοντα υπόψη το γεγονός ότι η ρύθμιση της ώρας είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, ε, τελικά τι θα συμβεί εάν οι προσπάθειες για εναρμόνιση ε, καταλήξουν σε διέξοδο, ίσως κάπου στη μέση. Κατά τη δική μου άποψη, αυτό είναι και ένα βασικό στοιχείο το οποίο κατά κάποιον τρόπο παρεμποδίζει και τις συζητήσεις στο Συμβούλιο. Υπάρχει πρόβλημα με αυτό το θέμα και δεν ξέρω ε, ποια θα ήταν η διέξοδος εάν κατά κάποιον τρόπο ε, προσκρούσουν οι διαπραγματεύσεις αδιέξοδο. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ντέλη, ο εισηγητή και εγώ είμαι εγγεγραμμένο στον κατάλογο των ομιλητών και θέλω να σα πω το εξή. Κοιτάξτε, στη Γερμανία η σημασία αυτού του θέματο ποτέ δεν είχε προβληθεί τόσο πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε επιτέλου κάντε κάτι, είναι υπέροχο και στηρίζουν αυτή την πρόταση και υπάρχουν οι άλλοι που λένε συγγνώμη δεν έχετε να κάνετε τίποτα καλύτερο από το να ασχολείστε με αυτό το αμεληταίο θέμα. Κάπου λοιπόν πρέπει να βρούμε μια λύση. Εγώ είμαι υπέρ τη κατάργηση τη αλλαγή ώρα γιατί εκνευρίζει πάρα πολύ. Και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο επ' αυτού. Έχουμε παρούσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Χάουκαρτ. Αν έχετε την καλοσύνη να μας πείτε και εσείς τη δική σας την άποψη. Θα είμαι σύντομος. Καταρχήν να ευχαριστήσω μία ακόμα φορά την εισηγήτρια, την κυρία Ούλσκοκ, και τους και εισηγητές για ε, την πολύ καλή δουλειά που έκαναν επί της πρότασής μας και στην πρόταση, το σχέδιο πρότασης. Είναι δύσκολο βέβαια να συντονιστούν τόσες επιτροπές, αλλά ήδη έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά. Καταρχήν να ευχαριστήσω την, την Επιτροπή σας για την συνολική της υποστήριξη στην πρόταση της Κομισιόν. Απαντώντας στην ε, ερώτηση του κ. Ρικέι, να σας υπενθυμίσω το πεδίο του Βελληνικές αυτής πρότασης. Προτείνει η Κομισιόν να εγκαταλείψουμε το σημερινό σύστημα όπου όλα τα κράτη-μέλη αλλάζουν ώρα δύο φορές το χρόνο, την ίδια στιγμή, την ίδια μέρα, με ένα πολύ εναρμονισμένο τρόπο και προτείνουμε να μετακινηθούμε σε ένα άλλο σύστημα όπου τα κράτη-μέλη θα καταργήσουν το ισχύον σύστημα ταυτόχρονα εναρμονισμένα και στο μέλλον θα αποφασίσουν να χρησιμοποιούν όποιο σύστημα επιλέξουν με εναρμονισμένο όμως τρόπο. Είναι δύσκολο αυτό. Αλλά Πιστεύω ότι και η κυρία Ουλσκοκ υποστηρίζει αυτή την πρόταση. Η Κομισιόν δεν σκοπεύει ούτε προτείνει να αναμειχθεί με την απόφαση του ποια ακριβώς ώρα θα έχει κάθε χώρα. Σε ποια ζώνη δηλαδή θα ενταχθεί. Είναι προφανές ότι κάθε κρατό μέλο έχει συμφέρον να ευθυγραμμιστεί με τους γειτονές του. Οπότε αυτό ισχύει πριν και πιστεύουμε αυτό θα ισχύει και στο μέλλον. Το σημαντικό είναι τα κράτη-μέλη να συντονίσουν τις επιλογές τους μεταξύ τους. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο μετάβασης από το σημερινό σύστημα στο επόμενο. Οπότε σημειώνουμε και κάποιες άλλες προτάσεις που έχουν γίνει. Για παράδειγμα, την σύσταση εθνικών σημείων επαφής ή το συντονισμό της, ε, ε, θέσεις και των επιλογών των κρατών μελών. Όμως αυτές οι επιλογές, αυτές οι θέσεις εξακολουθούν να είναι εθνική αρμοδιότητα και εντάσσονται στο πλαίσιο της επικορικότητας. Οπότε ας το σκεφτεί αυτό το Κοινοβούλιο όταν οριστικοποιήσει τη θέση του. Τώρα, για το θέμα ε, του πότε θα τεθεί σε ισχύ η οδηγία. Αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται λίγο περισσότερος χρόνος από ό,τι αυτό που είχαμε προτείνει αρχικά. Οπότε χρειάζεται να δώσουμε μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο έτσι ώστε όλοι οι πολίτες καθώς επίσης και οι αγρότες, οι επιχειρήσεις και ο κρατικός τομέας να βρουν τις κατάλληλες λύσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε την ψηφοφορία σας αρχές Μαρτίου και την υιοθέτηση αργότερα τον επόμενο μήνα στην Ολομέλεια. Η υιοθέτηση θέσεις από πλευράς του Κοινοβουλίου πριν διακοπούν οι ε, συνεδριάσεις σας πρώτων εκλογών θα είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα για το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ να ολοκληρώσω δίνοντας το λόγο στην κυρία Ουλουσκόκ έτσι ώστε να απαντήσει στις ερωτήσεις που ατέθησαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα επαναλάβω και εγώ αυτά που είπε ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να απαντήσω στον κύριο Βάντεκαμπ. Στην ε, Επιτροπή μας θα ψηφίσουμε στις 4 Μαρτίου. Στην Ολομέλεια θα ψηφίσουμε στα τέλη Μαρτίου και μετά θα περιμένουμε το Συμβούλιο. Θα εξαρτηθεί λοιπόν από το πότε θα καταλήξει το Συμβούλιο σε κάποια θέση, αλλά ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό ή στα τέλη του προσεχού ε, του, του σπουδιανίου ή του επόμενου, στις αρχές του επόμενου. θα επικοινωνήσουμε με το Συμβούλιο και θα του ζητήσουμε να θέσουν το θέμα αυτό ως προτεραιότητα και θα τους παροτρύνουμε λοιπόν να υιοθετήσουν ένα πιο φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτά που υπόθηκαν, σίγουρα θέλουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δείξουμε ότι αρκούμε τους πολίτες, ότι ασχολούμαστε με αυτούς και ενσκύπτουμε στα προβλήματά τους. Υπάρχουν ορισμένοι πολίτες που είναι περίπου κανένα δύο εκατομμύρια οι οποίοι θέλουν επιτέλους να γίνει κάτι με την εποχιακή αλλαγή ώρας. Υπάρχουν ορισμένοι που πιστεύουν πως δεν πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή διότι θα επηρεάσει την υγεία και την καθημερινότητα των πολιτών. Και ίσως ε, ορισμένοι θεωρούν πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα έπρεπε να ασχολείται με τέτοια θέματα, όμως είμαστε εδώ γιατί μας έχουν εκλέξει πολίτες περιμένουν από εμά να ασχοληθούμε με τα προβλήματά τους. Η εποχιακή αλλαγή ώρας ξεκίνησε με το σκεπτικό να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια της ενεργειακής ε, κρίσης. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα και είναι πιο δύσκολο και περίπλοκο να αλλάξεις κάτι και μάλιστα να τα αλλάζεις δύο φορές το χρόνο. Διότι σίγουρα έχει πολλές επιπτώσεις ψυχολογικά, βιολογικά. Δεν χρειάζεται να δραματοποιούμε την κατάσταση. Νομίζω πρέπει να φροντίσουμε η πρόταση να είναι σωστή. Δεν χρειάζεται να είναι επαναστατική, αλλά να είναι μια πρόταση που θα αντανακλά την άποψη των πολιτών ε, οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι ώστε να μην γίνεται αυτή η αιτήσια αλλαγή ώρας. Αυτό που πρέπει να αποφασίσουμε είναι αν θα παραμείνουμε μόνιμα στην ε, χειμερινή ώρα ή στη θερινή. Πραγματικά διαρωτώ με αν αυτή είναι τόσο δύσκολη και μεγάλη απόφαση για μας στο Κοινοβούλιο. δεν είναι τόσο σημαντικό το θέμα αυτό, αλλά για κάποιους ε, πολίτες όμως είναι πολύ σημαντικό να δουν ότι λαμβάνουμε αποφάσεις, ε, διότι έχουμε πέσει πολύ χαμηλά στα μάτια ορισμένων. Και πρέπει λοιπόν να έχουμε μία πρόταση, γι' αυτό λοιπόν σκοπεύουμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία, ε, ευχαριστώ πολύ, κυρία Ουλσκοκ για την ε, περίληψη που κάνατε. Σας ευχαριστώ. Να επαναλάβω αυτό που είπα και πιο πριν. Στην Επιτροπή Μεταφορών θα ψηφίσουμε στις 4 Μαρτίου και ελπίζω να ψηφίσουμε την έκθεση αυτή στην δεύτερη ολομέλεια του Μαρτίου. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα, Τελειώσαμε νωρίτερα. Έχουμε προγραμματίσει φωτογράφηση της Επιτροπής στις 11 και στη συνέχεια θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, οπότε θα διακόψουμε μέχρι τις 11. Να είστε εδώ στις 11 οι ευρωβουλευτές για τη φωτογράφηση.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 Après ce petit moment de détente et de... Μετά από αυτή τη μικρή διακοπή χαλάρωση και φωτογράφηση συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη. Allez, nous allons commencer, s'il vous plaît. Je suis heureuse. Με χαρά. Υποδεχόμαστε στην Επιτροπή μας τη νέα διευθύντρια, της, ε, εκτελεστική διευθύντρια τη ΕΜΣΑ, τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Θάλασσα, την κυρία Μάγια Μάρκοβιτσιτ Κόστελακ, που θα μα μιλήσει για την ΕΜΣΑ, την ε, συγχαίρω μία ακόμα γυναίκα, επικεφαλής ε, ε, Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1η Ιανουαρίου 2019. Ήδη έχουμε συνεργαστεί πολύ στενά με την ΕΜΣΑ και με τον προηγούμενο διευθυντή της, τον κύριο Μάρκου Μίλη. Εκτιμούμε πάρα πολύ την δουλειά, το έργο της ΕΜΣΑ, τις γνώσεις και την εξειδίκευσή της και τις παρεμβάσεις της στην Επιτροπή μας. Θα ακούσουμε δύο λόγια από εσά για το όραμά σας για την ΕΜΣΑ. Καλώς ήρθατε, η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή και σας δίνω το λόγο. Μετά θα συζητήσουμε με τους ευρωβουλευτές. Κύριε Βαντεκά, όλο μιλάτε σήμερα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, επτά μέλη της Ευρωβουλής, είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα για πρώτη φορά με το νέο μου, τα νέο μου τίτλο, τα νέα μου καθήκοντα της εκτελεστικής διευθύντριας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας στη Θάλασσα. Με τιμά η πρόσκλησή σας, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας το όραμά μου και τα σχέδιά μου για την ΕΜΣΑ. Έφτασα στην ε, υπηρεσία μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή. Έχουμε προκλήσεις αλλά και πάρα πολλές ευκαιρίες. Και ρόλος δικός μου είναι να εξασφαλίσω ότι η υπηρεσία θα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατό μπορεί τους πόρους που διαθέτει. Επιχειρησιακά να σας πω ότι ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ σημαντικός για την οικονομία μας. Πάνω από 80% του παγκόσμιου εμπορίου βασίζεται στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Οπότε εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ε, το 40% των συνολικών κόρων της παγκόσμιας ε, των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών ανήκουν σε ευρωπαϊκά συμφέροντα και τα λιμάνια μας είναι οι βασικές πύλες εισόδου. Συνεπώς και αυτά ε, γίνονται όλο και πιο σημαντικά όσο αυξάνεται το φορτίο που μεταφέρεται. Όλα βέβαια αλλάζουν. Έχουμε όλο και περισσότερα μεγαλύτερα σκάφη. Μερικά από αυτά φτάνουν σε μέγεθος τρία γήπεδα ποδοσφαίρου. Δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι η τεχνολογία και οι τεχνολογικές εξελίξεις ε, αλλάζουν την καθημερινότητά μας. Και εδώ αναφέρομαι πιο πολύ στις, στα αυτόνομα σκάφη. Είναι μια εξέλιξη η οποία βρίσκεται ήδη στο ραντάρ μας και είναι πιθανό να αλλάξει μια για πάντα τις θαλάσσιες μεταφορές όπως γνωρίζουμε σήμερα. Αυτή η, ό, όσο τη στιγμή που γίνεται αυτό αντιλαμβανόμαστε και τις επιπτώσεις της, ε, των θαλάσσιων μεταφορών στο περιβάλλον. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία για να μειώσουμε και το περιβαλλοντικό ίχνος των θαλάσσιων μεταφορών. Σύντομα θα εκλεγεί καινούργο κοινοβούλιο από θεσμικής πλευράς, καινούργια κομισιόν και αναμένουμε και το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2021. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή σας που έχει προτείνει να διατηρηθεί σταθερά ε, σταθερός ο προπολογισμό της υπηρεσίας μας και σε ονομαστική και σε πραγματική αξία. Λαμβάνοντα υπόψη και την ε, επιχειρησιακή και την θεσμική πτυχή, λοιπόν, υπόψη, λαμβάνουμε, ε, ετοιμάζουμε το καινούργιο μα ε, πρόγραμμα εργασιών, την καινούργια μα εργασία που θα υποβληθεί πριν το τέλο του χρόνου. Είναι σημαντική προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία τη υπηρεσία μα. Η στρατηγική αυτή θα είναι φιλόδοξη. Γι' αυτό είναι σημαντικό να την επεξεργαστούμε σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέρη, τα οποία εκπροσωπούνται στο Διοικητικό μας Συμβούλιο. Θα, η στρατηγική αυτή θα αναγνωρίζει την ΕΜΣΑ ως οργάνωση στην αιχμή της ε, τεχνολογικής εξέλιξης και ως κέντρο αριστείας για θέματα σχετικά με τη θάλασσα. Τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν οι βασικοί μας πελάτες. Και θα εξακολουθήσουμε να τους προσφέρουμε Τη υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Έτσι ώστε και αυτοί, κράτη-μέλη και κομισιόν, να ε, φέρουν σε πέρα τα δικά τους καθήκοντα. Ταυτόχρονα θα ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες και φορείς, προκειμένου να αυξήσουμε την προστιθέμενη αξία που προσφέρουμε στον τομέα των θαλάσσιων μεταφόρων. Επίσης, θέλω η ΕΜΣΑ να γίνει πιο ορατή σε διεθνές επίπεδο και ως εξαγωγέας ευρωπαϊκών λύσεων αλλά και, ο, και προβάλλοντας τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Για να γίνει αυτό θα βελτιώσουμε τις εσωτερικές μας διαδικασίες και θα τις ευθυγραμμίσουμε με τα διεθνή στάνταρ. Όλες οι υπηρεσίες μας έχουν ως στόχο την αύξηση της ασφάλειας θάλασσα και την προστασία του περιβάλλοντος καθώς επίσης και προετοιμασία έναντι ε, ε ατυχημάτων στη θάλασσα και μόλυνσης. Οι μελλοντικές προσπάθειες θα εστιαστούν στην ολοκλήρωση, την, ε, στην ένταξη στις εργασίες μας της παρακολούθησης της κατάστασης θάλασσας. Ε, είναι πολύ σημαντικό να συνδεθούμε και με τις διαδικασίες παρακολούθησης των ακτών. Ε, θέλουμε διάφορα επίπεδα με διάφορα δικαιώματα πρόσβασης στις υπηρεσίες μας. Ε, στηρίζουμε 3.300 χρήστες σε 240 διαφορετικές οργανώσεις. Και αυτά τα νούμερα αυξάνονται συνεχώς. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες μας γίνεται όλο και πιο φιλική προς το χρήστη με την καινούργια έκδοση της ε, εφαρμογή μας για κινητά τηλέφωνα, η οποία, για κινητές συσκευέ, η οποία δημοσιεύτηκε πέρσι. Ε, με τα δεδομένα που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας μπορούμε να εξερευνήσουμε περισσότερους τρόπους να τα εκμεταλλευτούμε. Πέρσι, για παράδειγμα, ξεκινήσαμε ε, το εργαλείο παρακολούθησης της αυτόματο, αυτόματης συμπεριφοράς είναι ένας αλγόριθμος, ένα εργαλείο που βασίζεται σε ένα αλγόριθμο που αναλύει τα δεδομένα θέσεις των πλοίων και ε, αυτοματώς εντοπίζει ύποπτες συμπεριφορές. Σε πραγματικό χρόνο μάλιστα μπορεί να σημάνει ε, τον κόδωνα του κινδύνου. Έχουμε πάνω από 400 χρήστες και πάνω από 2.000 τέτοιου είδους ειδοποίησης ε, ε, που έχουν σχέση με την αλληλεία, με την προστασία των συνόρων, ε, το περιβάλλον κλπ. Τα δεδομένα επίσης θέλουν να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για τη διαμόρφωση πολιτικών. Μία άλλη σχετικά καινούργια δραστηριότητα της ΕΜΣΑ που αναπτύχθηκε προκειμένου να συμπληρώσει την εικόνα που έχουμε για τη θάλασσα είναι οι υπηρεσίες ΑΡΠΑ. Από αυτό το slide βλέπετε ότι ήδη παρέχουμε ε, υπηρεσίες παρακολούθησης κατάστασης θάλασσα και μέσω αεροπλάνων. Ε, το 2018 ολοκληρώθηκε με μια δημοπράτηση που διευρύνει τις δυνατότητές μας. Έχουμε πλέον και καθέτο απογειώσεως αεροπλάνα και μικρότερα αεροπλάνα, τα μικρότερες συσκευές οι οποίες μπορούν να απογειωθούν από πλοία. Ήδη το συμβόλαιο έχει ε, δοθεί, ε, έχει κατακυρωθεί. Θα πρέπει κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες να ρυθμιστούν, αλλά η υπηρεσία μας είναι ήδη διαθέσιμη. Χρησιμοποιείται ήδη, για παράδειγμα στην Πορτογαλία και την Ισπανία και σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία στην Ισλανδία και στη δική μου χώρα την Κροατία. Μέχρι το τέλος του χρόνου προγραμματίζουμε υπηρεσίες ARPA να είναι διαθέσιμες στη Δανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Frontex και την ΕΦΚΑ. Η ΕΜΣΑ στηρίζει τη, τη διαδραστηριότητα της θάλασσα και από τη γη. Έχουμε το σύστημα εντοπισμού ε, των παράνομων εκφορτώσεων, καθώς επίσης και της μόλις στη θάλασσα. 5.000 περίπου εικόνες δόθηκαν το 2018, 30 λεπτά μετά την λήψη τους από το δορυφόρο. επι, ε, συνολικά προσφέρουμε εικόνες οι οποίες θα βοηθήσουν στην κατανόηση της κατάστασης και στη, και στη θάλασσα. Ε, η υπηρεσία αυτή είναι, διατε, διατίθεται για εγκεκριμένου χρήστες ε, που έχουν σχέση με την, τον έλεγχο της τελωνία, εφαρμογή του δικαίου, του, του νόμου, προστασία του περιβάλλοντος, θαλάσσια μόλυνση και ασφάλεια κλπ. Ο αριθμός των προϊόντων που προσφέρουμε και των υπηρεσιών μας αυξήθηκε κατά 40% πέρσι. Σήμερα πιο πολύ από ποτέ χρειάζεται όχι μόνο να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη τεχνολογίας, αλλά να την προλάβουμε κιόλας, να την προκαταβάλουμε. Γιατί η τεχνολογία μπορεί να φέρει επαναστατικές αλλαγές. Για παράδειγμα, αυτόνομη, αυτόνομα σκάφη. Ξεκινάμε λοιπόν μία μελέτη για την, ε, ε, τον αντίκτυπο της χρήσης αυτόματων, αυτοματοποιημένων σκαφών ε, παρακολούθησης. Θα μας επιτρέψει αυτή η μελέτη να δούμε πώς μπορούμε να εντάξουμε τέτοιου τύπου εξελίξεις στο δικό μας σύστημα. Η ΕΜΣΑ επίσης θα διερευνήσει πώς μπορεί να ωφεληθεί από υπηρεσίες στο υπολογιστικό νέφος. Οι ευκαιρίες που φέρνει αυτή η τεχνολογική ε, ε, αυτή η τεχνολογία ε, είναι τεράστιες. Πρόσφατα διοργανώσαμε ένα εργαστήριο στην ΕΜΣΑ με διάφορες άλλες υπηρεσίες, με την ΕΝΙΣΑ για παράδειγμα, προκειμένου να δημιουργήσουμε, να ε, χτίσουμε ε, ε, τύχη των απειλών που μπορεί να προκύψουν εξαιτία των υπηρεσιών που θα προσφέρονται στο νέφος, για παράδειγμα κυβερνοεπιθέσεις. Θέλουμε επίσης να προλάβουμε τη μόλις στη θάλασσα. Θα διερευνήσουμε πού, πώς μπορεί η ΕΜΣΑ να εμπλακεί περισσότερο και στην ανακύκλωση του έρματος των πλοίων. Ε, ε, θα εργαστούμε εξετάζοντας εναλλακτικά κάψιμα για τα πλοία. Στην πενταετή μας στρατηγική θέλουμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε και στην μείωση των εκπομπών ε, το, των εκπομπών, των απορρίψεων ε, οργανικών προϊόντων ε, και πλαστικών στη θάλασσα. Επίσης, στηρίζουμε τις παράκτιες χώρες για να αντιμετωπίζουν θέματα μόλις στη θάλασσα. Έχουμε 17 σκάφη αντιμετώπιση τέτοιων μολύνσεων, τα οποία είναι μοιρασμένα σε όλη την έκταση των θαλασσών μας. Ε, τα ενοικιάζουμε και συμπληρώνουν άλλου τύπου υπηρεσίες μας που αν προσφέρονται ανάλογα με τις ανάγκες. Ε, για παράδειγμα εξοπλισμό, απομόλυνσης, ε, με τρόπο που να έχουμε διάφορες δυνατότητες απόκρισης ανάλογα με τη μορφή της μόλυνσης. Πολύ συχνά εστιαζόμαστε στον ίδιο τον εξοπλισμό ξεχνώντας το ανθρώπινο δυναμικό. Η κοινωνική ατζέντα και το ανθρώπινος παράγοντας όμως θα πρέπει να παραμένουν στο επίκεντρό μας. Η υπηρεσία μα θα προσφέρει ε, μαθήματα επιμόρφωσης ε, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και στην τεχνολογία. Για παράδειγμα, η εικονική τεχνολογία, εικονική πραγματικότητα θα χρησιμοποιηθεί σε αυτά τα μαθήματα. Ε, θα προσπαθήσουμε να διευρύνουμε επίσης τους συμμετέχοντες και τα θέματα τα οποία θα καλύπτονται. Το 2019 ο IMO έχει ως ε, κεντρικό θέμα τις γυναίκες. Ε, Δεδομένου ότι η Επίτροπος είναι γυναίκα, δεδομένου ότι εγώ είμαι γυναίκα, δεδομένου ότι η Πρόεδρό σα είναι γυναίκα, μπορώ να σας ανακοινώσω ότι και η ΕΜΣΑ θα προβάλλει δραστήρια το θέμα των ίσων ευκαιριών στον τομέα της ναυτιλίας. Η ΕΜΣΑ έχει οριμάσει αρκετά και οι ικανότητές μας, οι δυνατότητές μας προσελκύουν το ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο. Ήδη προσφέρουμε τεχνική συνδρομή στι πολιτικέ γειτονίε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μα επιτρέπει να βελτιώσουμε συνολικότερα την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντο εντό των σύνορων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συχνά δεχόμαστε αντιπροσωπείες, επίσκεψη αντιπροσωπείων από τρίτε χώρε που προσπαθούν να ενημερωθούν. Εδώ βλέπω μια δυνατότητα η ΕΜΣΑ να εξάγει τις ευρωπαϊκές λύσεις και να προβάλλει τις πολιτικές μας διεθνώς. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που έχετε στηρίξει την, το έργο μας και θα ήθελα να σας, καλώσω, να σας ε, προσκαλέσω να μας επισκεφτείτε όπως κάνατε και πέρσι. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Madame la Présidente, euh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε της ΣΕΜΣΑ. Πολλά αυτά που μας είπατε. Μιλήσατε για τη μόλυνση, για τις νέες τεχνολογίες, για την κλιματική αλλαγή και για τις ε, δημοσιονομικές στρατηγικές. Θέλω να ανοίξω τη συζήτηση και θα ξεκινήσω με τον κύριο Φάντενκαμπ. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ε, θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά την κυρία Μάρκοβιτς Ίσως δεν προφέρω πολύ καλά το όνομά σας, ε, γιατί τα κροατικά μου ε, δεν είναι ακόμα καλά, αλλά διάβασα στο βιογραφικό σας ότι ασχοληθήκατε σε μια διατριβή ε, κυρίως με την ανακύκλωση του έρματος και αυτό είναι κάτι το πολύ συγκεκριμένο που αφορά τον κλάδο. Εγώ έχω μία άλλη ερώτηση. Η συνεργασία ανάμεσα στην ΕΜΖΑ, την Frontex και τον Οργανισμό Αλίας, τι γίνεται με αυτή τη συνεργασία, τι μορφή έχει λάβει. Κατόπιν, κάτι πολύ συγκεκριμένο, όσον αφορά την παράνομη διακίνηση ανθρώπινων όντων. Γνωρίζουμε όλοι ε, τις ε, δυσάρεστες αυτές ιστορίες ε, στη Μεσόγειο και πριν από κάποια χρόνια έθεσα αυτή την ερώτηση στους ε, προκατόχους σας. Ε, τώρα βλέπουμε ότι προκύπτει και ένα άλλο θέμα, ε, παράνομο εμπόριο στη Βόρειο Θάλασσα. Και θέλω να σας ρωτήσω, ε, πώς ακριβώς ε, κατανέμονται αυτές οι αρμοδιότητες άμεσα στους τρεις οργανισμούς που προανέφερα. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά τον IMO, τον Διεθνή Οργανισμό ναυτιλίας. Δεν αναφερθήκατε στο θέμα αυτό, αλλά εγώ είχα ακούσει ότι η ΕΜΖΑ ε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον οργανισμό IMO. Οφείλουμε λοιπόν ε, να δώσουμε κάποια κίνητρα σε αυτούς τους ε, απαράδεκτους τους Αμερικανούς οι οποίοι εξακολουθούν να μολύνουν τη θάλασσα και το περιβάλλον. Λοιπόν, θα συνεχίσω στα αγγλικά για να μην τα περιπλέξω περαιτέρω τα πράγματα. Όπως σας είπα, μήπως μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται με την έμψα, τη σχέση ανάμεσα στην έμψα και τον ΑΕΜΟ, την έμψα τη δική μας και τον ΑΕΜΟ και τι γίνεται ε, σχετικά με την συγκέντρωση δεδομένων για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τους εκλογείς αφορά τις πλαστικές ύλες, ε, την ε, μόλυνση των θαλασσών μας. Ε, δεν ξέρω ακριβώς, εσείς είστε επικεφαλής για τον καθαρισμό των θαλασσών, αλλά ποιος το, αν όχι ποιος το κάνει αυτό, είναι μια σκέτη απλή πρωτοβουλία ή εμπλέκεται και η ΕΜΣΑ. Θέλω λιγάκι να ρωτήσω για τα drones και για τους πρόσφυγες όταν ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος της ΕΜΖΑ βλέπει ένα σκάφος που βρίσκεται σε αναταραχή, τι ακριβώς κάνετε εκεί. Θεωρείτε ότι είναι δουλειά σα, παίρνετε τηλέφωνο τη Frontex, δεν κάνετε τίποτα. Τι ακριβώ κάνετε, θα ήθελα να γνωρίζω. Για να ανακεφαλαιώσω. Ποια είναι η συνεργασία ανάμεσα στην ΕΜΣΑ, τη Frontex και άλλου οργανισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, ποια είναι η σχέση με τον ε, Διεθνή Οργανισμό ε, Ναυτιλίας. Και τρίτη ερώτηση, πώ ακριβώ καθαρίζεται τις θάλασσές μας. Η κυρία Άντερσεν η επόμενη. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Πρόεδρε. Σας καλωσορίζουμε θερμά σε αυτή την Επιτροπή. Ε, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Όπως ξέρετε, αυτή η Επιτροπή έχει κάνει πολλή δουλειά για την ε, νομοθεσία για θέματα θαλασσών. Πρόσφατα, με μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώσαμε μία συμφωνία όπου καταλήξουμε ότι ε, θα εξετάσουμε περισσότερες λεπτομέρειες την εκπαίδευση των ναυτικών, την πιστοποίηση των επιτυχίων τους. Η ΕΜΣΑ παίζει εκεί ρόλο και θέλουμε να ρωτήσουμε ε, εσείς τι ακριβώς κάνετε για να αποκτήσουμε σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό ναυτικού που να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, και με ενδιαφέρει λοιπόν η αποψία για αυτή τη συμφωνία να μας πείτε επίσης μήπως μπορούμε να κάνουμε και και κάτι άλλο σε επιτροπή για να βοηθήσουμε την ΕΜΣΑ έτσι ώστε πράγματι να μπορέσουμε να καλύψουμε τις περισσότερες φιλοδοξίες ε, των ναυτικών μας. Παρεπιπτόντως υπάρχει και μια άλλη ε, ρήτρα που μιλάει για τα πτυχία των ναυτικών. Ε, θέλω να είμαστε σίγουροι ότι ό,τι κάνουμε σε αυτόν τον τομέα είναι απόλυτα συμβατό όχι μόνο με τους κανονισμούς για την εκπαίδευση των ναυτικών αλλά και με τις διατάξεις των ε, συνθήκων για τους ε, εργαζόμενους σε διεθνές επίπεδο. Θέλω οπωσδήποτε οι δικοί μας οι ναυτικοί και οι εκπαιδευόμενοι να καλύπτουν τα ανώτατα κριτήρια στο ανώτατο επίπεδο. Ε, εγώ χάρηκα πάρα πολύ με αυτή τη συμφωνία και πραγματικά προσβλέπω στην απάντησή σας. Πολύ ωραία. Η κυρία Φώστερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε και θα ήθελα να καλωσορίσω την επικεφαλής της ΕΜΣΑ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόσαστε εδώ σήμερα το πρωί. Ε, θέλω να αναφερθώ σε τρεις βασικούς ε, τομείς. Ένας εξ αυτών αναφέρθηκε είναι ο IMO. Ε, η ΕΜΣΑ είναι υποχρεωμένη προφανώς και να σέβεται όλους τους κανόνες και κανονισμού που έχουν θεσπιστεί εδώ και δεκαετίες. Δείτε λοιπόν το εξής ερώτημα. Εσείς πώς ακριβώς ασκείτε επιρροή μέσα σε αυτόν τον οργανισμό, των ΑΕΜΟ που είναι σχετικά νεόκοπος, ε, κατά την άποψή μου τα καταφέρνει αρκετά καλά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το δεύτερο θέμα έχει σχέση με τα drone. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ το θέμα αυτό, γιατί ήμουν εισηγήτρια για τα drone. Βέβαια, αυτά τα συνδέουμε κυρίως για τις ε, αερομεταφορές. Ε, ε, στο Λονδίνο. Υπάρχει εκεί ε, η εκπροσώπηση πολλών εταιριών που ασχολούνται με τα drones. Άρα δηλαδή αυτό που με ενδιαφέρει είναι το ότι τα drones από ό,τι βλέπετε τώρα ε, χρησιμοποιούνται και στις θάλασσες για να μπορείτε να παρακολουθήσετε τα μεγάλα σκάφη, τη συντήρησή τους. Δεν πρόκειται μόνο δηλαδή για γενικότερη ασαφή παρακολούθηση. Όλα αυτά σημαίνουν ότι θα πρέπει να υπάρχει και απαραίτητη τεχνογνωσία. Και έτσι φάνω, φτάνω σε αυτό που θέλω να καταλήξω, δηλαδή ε, είναι σημαντικό, ε, το δείξατε, και τα παιδιά στο σχολείο και όλοι παρακολουθούν ε, τα πλαστικά απόβλητα στις ε, θάλασσες. Ίσως λοιπόν και τα drones μπορούν εδώ να παίξουν κάποιο ρόλο. Αυτό όμως που με απασχολεί είναι το εξής. Ε, μπορούμε βέβαια όλοι να μιλάμε για το ποιο πρόγραμμα θα πειράσει... την χλωρίδα, την πανίδα, τα ψάρια. Αυτό το πρόβλημα αφορά όλο τον κόσμο και παίζει ρόλο ο ΑΕΜΟ. Μπορούμε βέβαια να θεσπίζουμε κανονισμούς, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τους κανονισμούς και τους κανόνες που θεσπίζουμε διότι αλλιώς αν δεν έχουμε μια διαδικασία εφαρμογής των μέτρων, αν δεν προβλέπονται πρόστιμα, αν δεν μπορούμε να αποτρέψουμε το να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, ε, τότε κατ' ουσίαν ναι μεν όλοι μιλάμε για το πόσο τραγικά είναι όλα αυτά, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Εσείς ως ΕΜΣΑ τι ακριβώς πρόγραμμα έχετε για να αντιμετωπιστεί αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία να έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια κυρία Μαρκοβίτς για την νέα ε, σας θέση. Χαιρόμαστε πολύ που βρίσκεστε εδώ. Φορέστε τώρα τα ακουστικά σας γιατί θα μιλήσω γερμανικά. Θεωρώ Πολύ ωραίο που είναι μια γυναίκα επικεφαλής της ΕΜΣΑ. Με τον ε, προκατοχό σας κύριο Μούλερ είχαμε πολύ καλή συνεργασία, όμως σαν γυναίκα χαίρομαι πάρα πολύ που έχω απέναντί μου μια γυναίκα. Και είπατε πως ε, θέλετε να δείτε ε, την ΕΜΣΑ να δίνει περισσότερες ε, ίσες ευκαιρίες. Μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυτό και στην ναυτιλία, να γίνει πιο ελκυστική για τις γυναίκες, διότι οι γυναίκες όταν σκέφτονται την ναυτιλία λένε «αυτό δεν είναι για μένα». Οπότε θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε, να προσπαθήσετε εσείς μάλλον να δώσετε μία έμφαση σε αυτό. Τώρα, τα έρμα είναι κάτι το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ. Αν γνωρίζετε, ήμουν ε, εισηγήτρια για την αναθεώρηση της ε, οδηγίας για τις υποδομές των λιμένων δεν καταφέραμε να περάσουμε ε, τις ε, αλλαγές που θέλαμε, τα κράτη-μέλη είχαν προβάλει αντίσταση και αυτό που περιμένουμε από την ΕΜΣΑ είναι να ασχοληθεί πολύ πιο έντονα με τις ε, εγκαταστάσεις υποδοχής τους λιμένες, διότι έχουμε όλη την πεποίθηση πως η δουλειά που κάνατε είναι πάρα πολύ καλή, αλλά το σημαντικό είναι οι θάλασσες να είναι καθαρές και θα πρέπει ο καθαρισμός των λιμένων να γίνεται με καλύτερο τρόπο και επίσης ε, να γίνεται καλύτερος έλεγχος των εργασιών. Ε, και πρέπει να αποφύγουμε αυτή την τακτική που τα πετάμε όλα στη θάλασσα και δεν τρέχει τίποτα. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ τουλάχιστον που έχετε αναφέρει κάτι τέτοιο, αλλά θα πρέπει να δούμε ε, μήπως μπορεί η ΕΜΣΑ να ε, αποκτήσει περισσότερες αρμοδιότητες ε, για τον τομέα αυτόν. Τώρα, Ο οργανισμός DLR επίσης που έχει έδρα στη Γερμανία θα μπορούσε να βοηθήσει σε ό,τι φορά τις δορφορικές επικοινωνίες. Ε, για να ε, εξετάσουμε την ε, δυνατότητα που έχουμε να χρησιμοποιήσουμε δορυφορικές επικοινωνίες για την ασφάλεια στη θάλασσα και τον καθαρισμό του βυθού. Στο Ευρωκοινοβούλιο από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διοργανωθεί μια εκδήλωση για το θέμα αυτό και ελπίζουμε η ΕΜΣΑ να συνεισφέρει σημαντικά. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει ε, εξεταστεί επαρκώς. Εδώ υπάρχουν πολλά που πρέπει να κάνουμε και η δική μας Επιτροπή έχει αναλάβει πρόσθετες αρμοδιότητες όπως και εσείς και όπως είπε ο κύριος ε, Μίλλερ, ο προκατοχός σας, ε, θέλουμε μία έμσα ικανοί, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ναι, θα τα καταφέρουμε, ξέρω πως ακούγεται έτσι κάπως περίεργα αυτό, αλλά ε, αυτό θα γίνει μόνο εάν αυξηθεί η χρηματοδότηση και το προσωπικό της ΕΜΣΑ. διότι χωρίς αυτό ε, η μία υπηρεσία δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της όταν αναλαμβάνει πρόσθετες αρμοδιότητες. Τώρα, όταν ήρθα σε εσά αυτό που ξέχασα να ρωτήσω είναι πού βρίσκεται το προσωπικό σας. Ε, είναι ε, προσωπικό που έχετε προσωπικο που ερχεται απο τη δίκηση, ε, εξωτερικό. Αυτό θα ήθελα να το μάθω. Και μετά, όταν μιλάτε για ενίσχυση του διεθνούς προφίλ, τι εννοείται ακριβώς. Εννοείται νέες διεθνείς επαφές, εννοείται προβολή περισσότερη, τι ακριβώς. Εννοείται πόσο πρέπει να τονίσουμε τον ε, τομέα της έρευνας, πώς μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε την εικόνα μας. Ο κύριος Τέιλορ. Ο κύριος έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε λοιπόν και συγχαρητήρια για τη νέα σας θέση. Είμαι σίγουρος πως θα τα πάτε περίφημα. Έχω τις εξής τρεις ερωτήσεις που μάλλον θα χρειαστούν περισσότερες, ε, περισσότερο για να απαντήσετε. Brexit καταρχάς. Τι σημαίνει το Brexit για την ΕΜΣΑ και πώς θα επηρεάσει τις υπηρεσίες που προσφέρει η ΕΜΣΑ στο Ηνωμένο Δεύτερη ερώτηση. Τον τελευταίο χρόνο σημειώθηκαν δύο περιστατικά ε, ενός μυστηριωδούς αερίου που ε, οδήγησε σε που στις νότιες ακτές της ε, Αγγλίας είχε οδηγήσει να πάνε πολλοί άνθρωποι στο νοσοκομείο. Μας είπατε πως δεν υπήρχε ο κατάλληλος εξοπλισμός για να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε ποιο αέριο ήταν αυτό και από πού προερχόταν. Όμως, η εξήγηση που δόθη, ε, η... μας είπατε μάλλον ότι ελπίζουμε τα drones να βοηθήσουν στο μέλλον σε αυτές τις περιπτώσεις. Πείτε μας περισσότερα γι' αυτό. Τέλος, το Κοινοβούλιο συμφώνησε με το ότι η ΕΜΣΑ θα είναι η αρμόδια υπηρεσία για τις ε, για την ασφάλεια στις ε, πλατφόρμες πετρελαίου και αερίου και για τον έλεγχο της ε, μόλυνσης. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μου πείτε πώς έχετε προχωρήσει σε αυτό το θέμα. Κυρία Αχνό, καλώς ήρθατε. Δεν θα επαναλάβω τις ερωτήσεις που έχουν ήδη λεχθεί. Με ενδιαφέρει συνεργασία με τη Frontex και ο, ο αντίκτυπος ε, της ε, μόλυνσης από τα πλαστικά. Ήδη ε, το, αναφέρθηκαν αυτές οι ερωτήσεις. Κύριε Κλούν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, καλή επιτυχία, κύριε Διευθύντρια. Η ναυτιλία έχει γίνει πολύ σημαντική πλέον με τις εξελίξεις εμπορικό, στον εμπορικό τομέα Το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου άλλωστε γίνεται μέσω των θαλασσών. Αναφερθήκατε στις ε, προκλήσεις που έχουμε στο μέλλον, επικοινωνία, μόλυνση, κλιματική αλλαγή, συνεργασία με τη Frontex και ε, τη Συνορφρουρά, πώς είναι αυτές οι σχέσεις, τι ρόλο παίζεται. Ε, έχουμε διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την ΕΜΣΑ, για παράδειγμα, ε, το ε, θέμα των διευκολύσεων στους λιμένες. Είναι λοιπόν ο ρόλος σας πολύ αναβαθμισμένος. Θα Ήθελα να μου πείτε ποια είναι η σχέση σας με άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες και οργανισμούς. Και τι θα γίνει αν η Βρετανία βγει τελικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στην θάλασσα της Ιρλανδίας. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι που ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ και για την ομιλία σας. Εσείς αναφερθήκατε στη βιωσιμότητα, παραπέμψατε σε νέες τεχνολογίες, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, τα ξέρουμε όλα αυτά. Όμως ε, για την πιο απλή εκδοχή εκεί δεν χρειάζεται να έχετε καμία τεχνολογική εξέλιξη. Ξέρετε ποιο θα ήταν να απαγορεύσετε το μαζούτ. Το μαζούτ ε, είναι κατ' ουσίαν προϊόν κατά κανόνα ή κανονικά το μαζούτ θα έπρεπε να χαρακτηρίζεται ως ειδικό απόβλητο. Δεν γίνεται όμως αυτό και τελικά τι γίνεται, φτάνει και σε εμά και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την κλιματική αλλαγή. Γι' αυτό λοιπόν το μαζούτ θα έπρεπε να είναι απαγορευμένο. Σε ορισμένε περιοχέ είναι απαγορευμένο, αλλά όχι παντού. Θέλω λοιπόν να σα πω, αν τελικά το μαζούτ αντικατασταθεί από το κανονικό δίζελ ε, το δίζελ έτσι κι αλλιώ και αυτό θεωρείται πολύ βρώμικο για του δρόμου Ευρώπη. Αλλά το μαζούτ, ε, αν μειωθεί κατά έστω 1%, ε, αυτό, θα αποδειχτεί ότι θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη ωφέλεια από τον ντίζελ. Γι' αυτό λοιπόν όταν πρόκειται για την προστασία του κλίματος, για τη Συμφωνία του Παρισιού, εσείς δεν τα λαμβάνετε όλα αυτά υπόψη σας. Μιλάμε ότι έχουμε ε, πηγές ε, που εκπέμπουν πολλές ουσίες επιβαρυντικές για το περιβάλλον. Εσείς τι πιστεύετε τι μπορεί να αλλάξει. Εγώ είμαι κάθετος να απαγορευτεί η χρήση μαζούτ γιατί οικονομικά ε, δεν θα είχε μεγάλες συνέπειες όμως οι προεκτάσεις ε, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε τους ε, πιο βρώμικους εκπομπής αερίων η Γκυζίνε ναι το ξέρει αυτό, το θίγουμε κάθε φορά το θέμα και ρωτώ εσάς, εσείς τι κάνετε, κανένα πρόβλημα, ε, συνεχίζουμε την πεπατημένη και περιμένουμε μέχρι να φτάσουμε στο υγροποιημένο αέριο που θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μετά από 20 χρόνια που και με συγχωρείτε και αυτό παρεμπιπτόντας θα είναι πάρα πολύ ακριβό. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στην κυρία Μάρκοβιτς Κώστελα. Πολλά έχετε να απαντήσετε, αλλά λίγο χρόνο. Έχετε το λόγο. Πολλές οι ερωτήσεις σας δείχνουν το ενδιαφέρον σας το, για το θέμα αυτό. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες, ομαδοποιώντας τις. Κάποιες ερωτήσεις είχαν σχέση με την, ε, τις υπηρεσίες που προσφέρουμε ε, για την ακτοφυλακή, ε, τη συνεργασία μας με την ακτοφυλακή. Όπως γνωρίζετε, έχει τροποποιηθεί ο κανονισμός που αφορά και μας και τη Frontex, προκειμένου να συμπεριληφθούν και αυτά τα καθήκοντα στην αποστολή μας. Αυτή η συνεργασία έχει ενταθεί 8 από τα καθήκοντα της ακτοφυλακής, ε, 6 ε, από τα 8 καθήκοντα της ακτοφυλακής ε, αποτελούν υπηρεσίες που προσφέρουμε εμείς. Οπότε πραγματικά βρισκόμαστε στο επίκεντρο της ανταλλαγής πληροφοριών για την ακτοφυλακή. Είμαστε δηλαδή ο οργανισμός που δίνει πληροφορίες σε όλα τα τελωνία και σε άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες, την Frontex, την, Frontex, την ΕΦΚΑ, αλλά και τις εθνικές υπηρεσίες που έχουν σχέση με την εκτοφυλακή. Εμείς έχουμε τις ολοκληρωμένες ε, θαλάσσιες υπηρεσίες, τις έχουμε αναπτύξει και συνεχίζουμε να τις αναπτύσσουμε, συλλέγουμε πληροφορίες και γι' αυτό το λόγο λειτουργούμε και με drones, γι' αυτό το λόγο θέλουμε να ανέβουμε και στο υπολογιστικό νέφος προκειμένου να διευρύνουμε το εύρος, το πλήθος των υπηρεσιών που προσφέρουμε χρησιμοποιώντας τη διαθέσιμη τεχνολογία. Θα τεθούμε επικεφαλής της συνεργασίας μας από φέτος και θα χορηγήσουμε περιβαλλοντική κατάρτιση σε όλους τους συμμετέχοντες στην συνεργασία σε θέματα ακτοφυλακής. Γιατί η ακτοφυλακή δεν έχει σχέση μόνο με την ασφάλεια, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με εμά την ΕΦΚΑ και την Frontex. Άλλωστε, σε αυτό συμμετέχουν και οι εθνικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε παρόντες στην Πορτογαλία, παράδειγμα, βοηθώντας την κυβέρνηση, τις εθνικές υπηρεσίες ε, και την Frontex. Έχουμε υπερτήσεις, οι οποίες συλλέγουν πληροφορίες, τις οποίες εμείς στέλνουμε στη Frontex και στην, στους κρατικούς φορείς, οι οποίοι έχουν ζητήσει την συνδρομή μας. Σε διεθνές επίπεδο ο IMO είναι η βασική παγκόσμια οργάνωση για θέματα θαλασσών και εμείς συμμετέχουμε στις εργασίες του ως τμήμα μέλος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής της Κομισιόν. Εκεί προβάλλουμε τις ευρωπαϊκές προτάσεις, ενημερωνόμαστε, συνεργαζόμαστε, οπότε είμαστε ήδη παρόντες στον IMO. Μπορούμε να είμαστε στο μέλλον ακόμα πιο δραστήριοι. Πώς? Παρέχοντας τεχνική συνδρομή μέσω του προγράμματος τεχνικής συνεργασίας που προσφέρεται από τον IMO στις αναπτυσσόμενες χώρες, σε αναπτυσσόμενες χώρες σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω ότι η Κομισιόν θα με στηρίξει. Έχουμε εντοπίσει τις περιοχές σε όλο τον κόσμο όπου τα ευρωπαϊκά συμφέροντα είναι πιο έντονα. Οπότε εκεί μπορούμε να προσφέρουμε αυτή την τεχνική συνδρομή προβάλλοντας τις δικές μας λύσεις ε, και εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Θα διασφαλίσουμε έτσι ότι οι ευρωπαϊκές λύσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας, θα γίνουν γνωστές σε όλο τον κόσμο. Εκεί βλέπω ένα ρόλο της ΕΜΣΑ εντός του IMO. Θα ήθελα επίσης η ΕΜΣΑ να συμμετάσχει πιο δυναμικά στη συνεργασία και με άλλους διεθνείς φορείς που έχουν σχέση με την αυτιλία και τη θάλασσα. Για παράδειγμα τον ILO, Έγινε μια ερώτηση για τους Ευρωπαίους ναυτικούς και σας ε, συγχαίρω για τη συμφωνία που πετύχατε ε, για την τροπολο... επί των τροπολογιών στην Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ο ILO έχει και άλλα εργαλεία, συμβάσεις μέσω των οποίων η ΕΜΣΑ μπορεί να βοηθήσει, για παράδειγμα, προσφέροντας εκπαίδευση προς τα, τις κυβερνήσεις. Έχουμε μπει σε μια νέα εποχή σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, ε, στην ΕΜΣΑ ετοιμαζόμαστε για την εικονική πραγματικότητα, ε, για τη χρήση, με τη χρήση προσωμιωτών και πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ τους ναυτικούς στην εκπαίδευσή τους. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο στο οποίο θα εργαστούμε είναι η αναβάθμιση του επαγγέλματος του ναυτικού. Μαζί με την Κομισιόν έχουμε ξεκινήσει μια, θα ξεκινήσουμε μάλλον μια καμπάνια, μια εκστρατεία για την πρόθεση του επαγγέλματος. Τώρα σε ό,τι αφορά τα πλαστικά, στην κοινωνία στρατηγική, όπως είπα, θα εξετάσουμε τις δυνατότητες η ΕΜΣΑ να συμμετάσχει περισσότερο και στην πρόληψη, γιατί εγώ είμαι πολύ υπέρ της πρόληψης, αλλά και στην καταπολέμηση του φαινομένου, την επίλυση του προβλήματος. Ε, εκεί εμείς μπορούμε να συνεισφέρουμε με τις πληροφορίες που μπορούμε να παράσχουμε, τις φωτογραφίες, τις εικόνες που συλλέγουμε, προκειμένου να μειωθεί η πίεση των πλαστικών υλών στο περιβάλλον. Δεν είναι εύκολο από τεχνολογικής πλευράς. Έχω μάθει ότι τα μικροπλαστικά δεν εντοπίζονται εύκολα από ένα αέρια μέσα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί καινούρια τεχνολογία. Έχω συζητήσει με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε τη χρήση των πλαστικών πάνω στα σκάφη. Μην ξεχνάτε ότι η ΕΜΣΑ ασχολείται κυρίως με την μόλις προέρχεται από τα ίδια τα σκάφη στη θάλασσα και όχι από πηγές που βρίσκονται στη στεριά. Οπότε είναι σημαντικό να μειώσουμε τη χρήση των πλαστικών πάνω στα σκάφη. Είναι ένας ε, μία από τις οδούς πρόληψης που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Τώρα, ε, τα drones, τα μη παντρωμένα αεροσκάφη αναφέρθηκαν πάρα πολλές φορές ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις διάσωσης. Θέλω να πω ότι οι δραστηριότητες που αναπτύσσουν τα drone, αυτό πρέπει να το αποφασίσουν τα κράτη-μέλη ή οι αρμόδιοι φορείς. Εμείς στέλνουμε τις φωτογραφίες ε, σε εκείνους που είναι κατ' ουσίαν αρμόδιοι στο να αναπτύξουν μια επιχείρηση επιτόπου. Ε, κατά κανόνα αρμόδιες είναι οι εθνικές αρχές. Ε, είναι κυρίαρχο δικαίωμά τους, είναι υποχρέωσή τους. Δηλαδή ε, βασικά εμείς τους στέλνουμε τις πληροφορίες και επίσης ε, βοηθάμε πολλές επιχειρήσεις διάσωσης και πάλι στα κράτη-μέλη προσφέροντας τις απαραίτητες πληροφορίες αλλά και την τεχνογνωσία για τεχνικά θέματα. Τα κυρίως μεγάλα, μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα πολύ μεγάλα, αυτές οι μεγάλες ε, μηχανές, αυτά βέβαια έχουν και τα αποκαλούμενα sniffers, ε, αυτές ε, τις συσκευές ε, που συγκεντρώνουν τις πληροφορίες από τα σκάφη. Ίσες ευκαιρίες και εκεί ετέθη ένα ερώτημα ή αν θέλετε μία παρατήρηση. Όπως σας είπα, αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα εξετάσουμε όχι μόνο στη στρατηγική μας, αλλά και στο πρόγραμμα δράσης μας. Θα καθορίσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές για τον τομέα της ε, ναυτιλίας, για τις θάλασσες. Δυστυχώς ε, στην πραγματικότητα, στην πραγματική θαλάσσια πολιτική δεν συμμετέχουν πολλές γυναίκες. Εμείς ε, προετοιμάζουμε ε, τα soft tools και το υλικό προβολής έτσι ώστε να συμμετέχουν περισσότερες γυναίκες στο μέλλον. Στη δική μας τη διοίκηση, στην ΕΜΣΑ, είμαστε κατά αναλογία 3 προς δύο. Δηλαδή ε, τρεις γυναίκες και δύο άνδρες. Εκεί έχουμε την πλειοψηφία. Πολύ καλό σε εμά. Βλέπετε σε εμά ισχύουν ίσε ευκαιρίε. Νομίζω η κυρία Πλούμ αναφέρθηκε στις ε, εγκαταστάσεις ελιμενισμού των σκαφών. Πράγματι, ήδη έχουμε λάβει μία εντολή στο να διασφαλίσουμε εναρμονισμένη εφαρμογή ε, δυνατοτήτων ελιμενισμού στα κράτη-μέλη. Επίσης ε, και οι αρμόδιοι για το περιβάλλον έχουν αναφερθεί στο θέμα αυτό. Είπατε και για την διαχείριση του νερού έρματος ε, σχετικά με τις εγκαταστάσεις ελιμενισμού. Υπάρχει όμως και το άλλο και στα σκάφη πρέπει να υπάρχει κάποια τέτοια πρόβλεψη. Στα λιμάνια το κόστος υποδοχής των νερών ε, έρματος ε, είναι πολύ ψηλό. Ε, λίγα κράτη διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα. Σε αυτό το τομέα έχουμε πολλά να κάνουμε για το νερό του έρματος και όσον αφορά τα σκάφη και όσον αφορά τον έλεγχο. Εμείς συμμετέχουμε στην εκπόνηση οδηγιών για το πώς θα ελέγχονται τα λιμάνια και αυτό είναι ένα εργαλείο το πώς μπορεί να, που μπορεί να διασφαλίσει την εναρμόνιση στους ε, κανόνες. Ε, πρέπει βεβαίως να υπάρχει και ο απαραίτητος εξοπλισμός πάνω στα σκάφη ε, και παρόλα αυτά υπάρχει α, ανασφάλεια κατά πόσον θα εφαρμόζονται οι κανόνες. Κατά τα άλλα, θέλω να αναφερθώ στο πρόγραμμα Κοπέρνικους. Προσπαθούμε να βελτιωθούμε μέσω αυτού. Και έχουμε και άλλα μέσα στη διάθεσή μας, γιατί αυτά είναι πολύ σημαντικά για την εικόνα μας. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα drone μεγάλων αποστάσεων χωρίς να έχουμε μία δορυφορική εικόνα πρέπει να έχουμε τους απαραίτητους δορυφόρους και γι' αυτό θέλω και να σας συγχαρώ για την πολύ σοφή ε, πολιτική απόφαση που λάβατε για την Ευρωπαϊκή Ενιαία Θηρίδα. Το θέμα αυτό ε, ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Εμείς θα προχωρήσουμε στις ε, τεχνικές λεπτομέρειες χρησιμοποιώντας και την δορυφορική τεχνολογία η οποία είναι απαραίτητη για να γίνεται πιο εύκολη καταγραφή ε, των ε, κανόνων που πρέπει να ισχύουν πάνω στα σκάφη. Όσον αφορά το προσωπικό, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι εμείς ε, έχουμε εμπειρογνώμονες πολύ εξειδικευμένου, τουλάχιστον κάτω από το πρίσμα των θαλάσσιων γνώσεων και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας που είναι να βοηθάμε τόσο την Επιτροπή όσο και τα κράτη-μέλη στην ανάπτυξη και στην παρακολούθηση περισσότερο της πολύπλοκης και περίπλοκης νομοθεσίας και σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο. Έχουμε βέβαια και πολλούς ε, εξειδικευμένους ηλεκτρονικούς γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτόν τον τομέα. Προσφέρουμε πολλές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Γι' αυτό λοιπόν ε, στο τον τομέα αυτό προφανώς και στηρίζουμε την ψηφιακή λύση. Αυτό που θέλω να δω κατά τα επόμενα πέντε έτη είναι και πλήρης ψηφιοποίηση των εσωτερικών μας διαδικασιών, ε, κάτι που δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι στο μέλλον δεν θα μιλάνε, θα συνεχίσουν να μιλάνε, αλλά θα στέλνουν και mail και η χρήση της τεχνολογίας θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο την αποτελεσματικότητά μας. Όσον αφορά το Brexit, κάναμε αυτό που έχουν κάνει όλοι οι φορείς, δηλαδή έχουμε προετοιμαστεί για όλες τις δυνατές εξελίξεις. Βεβαίως δεν χαράσουμε εμείς πολιτικοί. Όμως εμείς ε, έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε οι δυνατόν να μειώσουμε ή ακόμα και να εξουδετερώσουμε οποιασδήποτε αρνητικές επιπτώσεις ε, στην ασφάλεια και στο περιβάλλον. η απαγόρευση χρήσης του μαζούτ. Μακάρι να γινόταν αυτό. Αυτό βέβαια είναι η προσωπική μου άποψη. Εγώ δεν είμαι πολιτικός, εσείς χαράσετε πολιτική. Πάντως να σας πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά για να περάσουν τα τελευταία χρόνια σε εναλλακτικά καύσιμα και θα πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι η ναυτιλία είναι ένας κλάδος που αναπτύσσεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν μπορούμε εμείς ε, να πηγαίνουμε αντίθετα από το ρεύμα. Αυτό θα καταστρέψει την ανταγωνιστικότητά μας. Όμως μπορούμε και εμείς να προβάλλουμε τις βέλτιστες λύσεις και αυτό κάνουμε μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, των κρατών μελών και του IMO. Πέρυσι ο IMO ε, έχει να επιδείξει αρκετές επιτυχίες και το Μάιο θα γίνει ένα βήμα περαιτέρω προς τον ε, καθορισμό του προγράμματος ε, δράσης. Παράλληλα, τόσο ο κλάδος όσο και οι ε, αρμόδιοι για την τεχνολογία αναζητούν τεχνικές λύσεις για να καταλήξουν στο ποια καύσιμα είναι και τα καλύτερα και για ποιο κλάδο του εμπορίου. Έχουμε ήδη σκάφη που κινούνται με υγροποιημένο φυσικό αέριο. Γνωρίζουμε όμως ότι αυτό δεν είναι η καλύτερη λύση γιατί ε, το LNG ε, έχει άλλες εκπομπές, όχι τόσο διοξίδιο του άνθρακα, αλλά οξίδια του αζότου, παραδείγματος χάρη. Θέλουμε να δούμε τι θα γίνει και με το υδρογόνο. Μόλις ε, τελικά οριστικοποιηθεί η τεχνολογία χρήσης υδρογόνου και έτσι θα είναι πολύ πιο εύκολο να απαγορεύσουμε τη χρήση μαζούτ. Ελπίζω να έδωσα ικανοποιητικές απαντήσεις. Αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, παρακαλώ είμαι στη διάθεσή σας. Ναι, ήσασταν πολύ ακριβείς και ευχαριστώ πολύ που απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ επίσης που ήρθατε να μας δείτε. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ΕΜΣΑ και να ξέρετε ότι θα είστε πάντα ευπρόσδεκτοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε και μια πολύ νέα ευρωβουλευτή εδώ που ήταν πολύ ισχύ σήμερα. Πώς σε λένε, πώς είναι το όνομά σου. Άνοιξε το μικρόφωνο. Τόνιτσκα. Χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς η πρόεδρος. <laughs> Όλοι για σένα εργαζόμαστε και για το μέλλον σου. Καλώς ήρθες. Τι Συνεχίζουμε. Ε, και κλεισμένων το θυρών για τους τριλόγους, για τους τριμές διαλόγους. Και το απόγευμα έχουμε συνάντηση των ε, συντονιστών. Παρακαλώ πολύ να σταματήσουμε το web streaming και ό.